Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε εδώ αυτούς που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οπότε, σας παρακαλώ, καθίστε πρώτα απ' όλα. Και πριν ξεκινήσουμε, έχω να κάνω κάποιες σημαντικές ε, ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι η συνάντηση αυτή περνάει στον ιστοχώρο όπως συμβαίνει και με άλλε συνεδριάσεις και θα συμβεί και τις επόμενες ε, τρεις μέρες που συνεδριάζουμε και ας είμαστε σε άλλη αίθουσα. Οπότε σας ζητούν οι υπηρεσίες να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο που βρίσκεται στα αριστερά σας γιατί συνδυάζεται με την ε, κάμερα που τραβάει και την εικόνα σας εκείνη τη στιγμή όταν παίρνετε το λόγο. Το εξαριστερόν σας μικρόφωνο λοιπόν να χρησιμοποιείτε. Εντάξει. Ωραία. Α, δεν έχετε. εντάξει, τότε πρέπει να ρωτήσουμε, να δούμε. Καθηνά να πούμε, όταν μιλάει στο γραφείο, τι στη χρησιμοποιεί. Καλά, εντάξει, ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή. Εγώ σας διαβάζω ότι οι οδηγίες μου δώσανε. Για την ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έπειτα, δυστυχώς η κυρία Χέντ δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα γενικά με τις μετακινήσεις, πάντως εκείνη είπε ότι σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε βγαίνει από την ημερήσια διάταξη η εκθεσή τη, αφού δεν είναι εδώ για να μα την παρουσιάσει. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί ένα ισχυώδη, αν μη του άλλο, φρόντισε να έρθει εδώ παρά τι δυσκολίε που είχε τι να κάνουμε. Ίσως στα διάφορα Τετάρτη το βράδυ, αν προλάβουμε, θα δούμε. Εντάξει με την ημερήσια διάταξη καταρχήν λοιπόν. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις. Πρακτικά των συνεδριάσεων της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου του 2009. Μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι, αν έχετε τίποτα αλλαγές να προτείνετε, να μας τις πείτε. Αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Και τώρα, περνάμε στο κυρίω θέμα που έχουμε σήμερα το απόγευμα. Μετά λοιπόν από πολλές ε, αλλαγέ, καθυστερήσεις, Ξαναρχίζουμε, ξαναβρισκόμαστε σε μια συνεδρίαση μαζί. Αύριο έχουμε και συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και μία πρώτη βίντεο διάσκεψη με την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ελπίζω να είσαστε όλοι και να έρθουν κι άλλοι, να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους παρόντες. Αλλά, στο μεταξύ, σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Η συγκήτρια είναι η κυρία Σάλντεμόζ. Οι περισσότεροι σκιώδες είναι εδώ, η κυρία Μακάρθιν δεν είναι, γιατί είναι άρρωστη σήμερα και θα την αντικαταστήσω εγώ. Η κυρία Κασταμπίλτης είναι εδώ, Κρότσμαν επίσης. Α, όχι, δεν είναι. Θα αργήσει. Εντάξει. Τέρναν,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 Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι λάβαμε την αγγλική μετάφραση όλων των τροπολογιών την Παρασκευή. Παρασκευή απόγευμα. Έχουμε λάβει 200 τροπολογίες πέρα από τις 80 που είχα εκπονήσει εγώ στη δική μου έκθεση. Γι' αυτό δεν ήταν δυνατό να εξετάσω αναλυτικά όλες τις τροπολογίες και να πάρω θέση. Θα ήθελα όμως καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για το μεγάλο τους ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Και εγώ βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα βρούμε συμβιβασμούς σε διάφορους τομείς. Αν και με την πρώτη ματιά φαίνεται να διήστανται αρκετά οι απόψεις μας ε, για κάποια από τα θέματα. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τα θέματα όπου πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμούς. Και θα ήθελα να καλέσω και τους σκιώδεις εισηγητές να μιλήσουν περισσότερο εις βάθος ε, για τις τροπολογίες τους. Ε, Πρωτού να μπω στα θέματα επί της ουσίας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων των συναδέλφων ότι Έχω συγκαλέσει δύο συναντήσεις σχεδόν εισηγητών τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ευτυχώς λοιπόν θα έχουμε χρόνο να εξετάσουμε αναλυτικά τα θέματα. Ας, κάνουμε, έχουμε λοιπόν μια πιο γενική συζήτηση σήμερα. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε με μονοσήματο τρόπο προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει η πρόταση αυτή. Δική μου επιθυμία ήταν τα αλκοολούχα να καλύπτονται από τον κανονισμό για τα τρόφιμα. Έχω ωστόσο την εντύπωση και δεν με εκπλήσει αυτό ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θέλουν τα αλκοολούχα να εξαιρούνται από τον κανονισμό για τα τρόφιμα. Γίνονται συζητήσεις ε, για το κατά πόσο θα πρέπει να εξαιρείται μόνο ο ίνος ή όλα τα αλκοολούχα ποτά. Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ κάποιων εξαιρέσεων και θα πρέπει να τις εξετάσουμε. Προσωπικά, εγώ θα ήθελα να συμπεριληφθούν οι κανόνες για τα αλκοολούχα. Μια... Ένα από τα άλλα θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το πού στη συσκευασία θα πρέπει να τυπώνονται οι πληροφορίες. Και εδώ έχουμε λάβει μια σειρά τροπολογιών, οι οποίες θέλουν οι πληροφορίες να μπαίνουν ή μπροστά στο πακέτο ή στην πίσω μεριά ή να μην υπάρχουν καθόλου κανόνες για το πού στο πακέτο θα πρέπει να τυπώνονται οι πληροφορίες. Εγώ θέλω μία λύση όπου οι πληροφορίες να πρέπει να αναγράφονται στο πακέτο με τρόπο ορατό και κατανοητό για τους καταναλωτές. Ε, δεν είναι απαραίτητο να είναι στο προστινό μέρος της συσκευασία. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε ο καταναλωτής να μην πρέπει να ψάξει ε, σε πολλά σημεία για να βρει τις ε, σχετικές πληροφορίες. Βλέπω επίσης ότι μια σειρά τροπολογιών έχει να κάνει με το μέγεθος του φόντου, το μέγεθος των γραμμάτων του κειμένου. Εγώ ε, μένω στην, ε, στο συμβιβασμό που, όπου καταλήξαμε στην προηγούμενη θητεία. Μερικοί θέλουν μεγαλύτερα γράμματα, άλλοι δεν θέλουν ε, συγκεκριμένες απαιτήσει για το μέγεθος των γραμμάτων. Και εδώ θα πρέπει να βρούμε κάποιον συμβιβασμό. Κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί απλά να γράφουμε ότι πρέπει να είναι ευαναγνωστό το κείμενο. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιγράψουμε και τι εννοούμε όταν λέμε ευανάγνωστο. Πιστεύω όμως ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση και για το θέμα αυτό. Με το θέμα αυτό συνδέεται και το εξής. Μια σειρά συναδέρφων ζητούν εξαίρεση ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασίας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ε, εξαιρέσει στο κατά πόσο καλύπτονται από την νομοθεσία. Και εδώ το φάσμα των απόψεων είναι πολύ ευρύ. Θα πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Η θέση μου είναι πάντω ότι γενικά θα πρέπει να προσέξουμε να μην συμπεριλάβουμε υπερβολικά πολλέ εξαιρέσει, διότι τελικά μόνο η μεγάλη παραγωγή θα καλύπτονται και τα πιο ε, σημαντικά προϊόντα θα καλύπτονται, αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε κάποιες λύσεις, ε, για παράδειγμα για τις συσκευασίε τσίχλας, ε, διότι είναι πολύ μικρές, οπότε είναι πολύ δύσκολο να, ε, συμπεριλαμβάνουν, να συμπεριλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες πάνω στη συσκευασία. Ένα θέμα που επίσης βλέπουμε σε πολλές τροπολογίες είναι το περιεχόμενο της δήλωση των διατροφικών πληροφοριών. Τι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό και τι θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε εδώ να βρούμε λύση ακούστηκαν επιθυμίες να ε, ε, ε, συμπεριλαμβάνουμε πληροφορίες για τις πρωτεΐνες, την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, άλατα κτλ. Εγώ νομίζω ότι ωφελεί τους καταναλωτές να γνωρίζουν τι περιέχεται μέσα στο προϊόν βασικά. Φυσικά θα έχουμε συζήτηση σχετικά με το πώς θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τα συστατικά ενός ε, τροφίμου. Προτείνεται ένα σύστημα ε, χρωματικών κωδίκων. Ε, κάποιοι συνάδελφοι συμφώνησαν με αυτό, όχι πάρα πολύ. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση που να δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ε, λαμβάνουν τι πληροφορίε που πρέπει και που να είναι και ε, λογική για τους παραγωγούς. Γενικά υπάρχει και μια συζήτηση για τις εξαιρέσεις γενικά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν ειδικού κανόνες στον τομέα αυτών. Θα πρέπει να δεχτούμε άλλες πληροφορίες από αυτές ε, που περιλαμβάνονται στο, στην Ομοθεσία περιτροφίμων. Μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν προαιρετικές ρυθμίσεις. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, διότι και εδώ έχουμε μεγάλο φάσμα απόψεων. Μερικοί θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίσουν δικούς τους κανόνες ε, παράλληλα με τον κανονισμό αυτό, ενώ άλλοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει κάτι τέτοιο να είναι δυνατόν. Για να μην σπαταλήσουμε τις προσπάθειές μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις ε, τις, διαφορές στην οτροπία που υπάρχουν ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Επίσης, έχει γίνει συζήτηση σχετικά με τη χώρα προέλευσης. Εγώ διστάζω σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματο αυτού, διότι πιστεύω ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει από πού προέρχεται το προϊόν του. Από την άλλη, θα πρέπει η λύση να είναι σκόπιμη, εφαρμόσιμη, να μην πρέπει οι παραγωγοί να αλλάζουν συσκευασίες και επίσης να μην καταλήξουμε σε προτεξιονισμό, σε προστατευτισμό. Η κυρία Μπίλτ υπέβαλε πρόταση η χώρα προέλευσης να ισχύει μόνο για τα βασικά τρόφιμα, τα κρέατα και τα ψάρια. Ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να το διευρύνουμε αυτό ώστε να καλύψουμε περισσότερε ομάδε προϊόντων. Να δούμε όμω μήπω μπορέσουμε και εδώ να βρούμε κάποιε λύσει. Να πω επίση ε, ότι υπά... ευτυχώ υπάρχουν και κάποια εύκολα θέματα εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφο που να διαφωνεί με την... τι υποχρεωτικέ απαιτήσει περί, ε, περί του ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να δίδονται ανά 100 γραμμάρια. Ε, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το, τα μεγέθη μερίδας ε, και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Άλλος τομέας ε, στον οποίο βλέπω να υπάρχουν εύκολες λύσεις για συμβιβασμούς είναι το θέμα για τις εξαιρέσεις για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Θα, θα ξαναπροσπαθήσω. Ένας ε, τομέας όπου πιστεύω ότι θα είναι εύκολο να βρούμε λύσεις θα είναι για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Δεν ξέρω πόσο γενικές θα πρέπει να είναι οι εξαιρέσει αυτές. Βλέπω όμως ότι αρκετοί συνάδελφοι θέλουν να ληφθούν υπόψη εδώ πέρα διάφορες ε, συνθήκες. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε πάλι να μην διευρύνουμε τόσο το πεδίο των εξαιρέσεων ώστε τελικά να καταλήξουμε να μην καλύπτεται τίποτα από την νομοθεσία. Επίσης, όσον αφορά τους κανόνες ε, για την επισήμανση που αφορά της αλλεργίας για τα μη προσκευασμένα τρόφιμα, θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση, η θέση μας είναι παρόμοια. Θα πρέπει ο καταναλωτή να λαμβάνει πληροφορίε σχετικά με αλλεργιογόνε ουσίε στα τρόφιμα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι διάφορε παραδόσει και νομοθεσίε στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θα μπω σε πολλέ ακόμα λεπτομέρειες. Παρακαλώ να μου παρουσιάσετε τις δικές σας τροπολογίες. Ένα τελευταίο θέμα θα ήθελα να θίξω, διότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες που λάβαμε αφορούν ε, θέματα που ήδη συζητήσαμε. Λάβαμε όμως και μία νέα πρόταση από τον Ούλε Σμιτ που προτείνει ε, να υπάρχει απέτηση για γραφή για τυφλούς στα τρόφιμα. Βρίσκω πολύ ωραία την ιδέα να βοηθήσουμε τους ε, τυφλούς συμπολίτες μας, αλλά θέλει το θέμα κατά πόσο είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είναι νέα η πρόταση αυτή, να ακούσω τις θέσεις σας. Ε, όπως είπα όμως, ε, χαίρομαι που ενδιαφέρεστε τόσο για το θέμα αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμούς, αν όχι για όλα τα θέματα, τουλάχιστον για κάποιες από τις πτυχές της πρότασης αυτής. Να πω όμως ότι είναι και απαραίτητο όλοι να δείξουμε κάποια ευελιξία για να καταλήξουμε σε κάποιους ε, συμβιβασμούς για να έχουμε μια ε, σωστή έκθεση τελικά, διότι οι απόψεις διήστανται αρκετά. Ε, θα κλείσω εδώ και περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μόζο, για τόσο τόσο ξεκάθαρα μας είπατε. Πράγματι, δεν θα ήταν και εύκολο να επεξεργαστείτε 280 τροπολογίες. Σίγουρα χρειάστηκε καλή συνεργασία με τους εισηγητές. Η κυρία Κράτσαμπλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Κρίστελ και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι προχωρήσαμε πολύ. Κάναμε πολλές προσπάθειες όλοι μας για να βρεθούμε πιο κοντά ένα στον άλλο, να προσεγγίσουμε τις απόψεις μας για το θέμα της προέλευσης, ε, της αναγνωσιμότητας των συσκευασιών και για τα 100 γραμμάρια της μερίδες και τα αλλεργογόνα συστατικά και το θέμα του κώδικα, αυτό που λέγαμε με σαν είναι το φανάρι της κυκλοφορίας με το κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε καταφέρει. Όμως ας με αφήσει η γραμματεία να μπορέσω να μιλήσω στον πρόεδρο και να με ακούει ο πρόεδρος. Έλεγα λοιπόν ότι όσον αφορά το ΕΛΚ, για τις ετικέτες στα προϊόντα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει τον ε, καταναλωτή, τον βοηθάει να κάνει όντας ενημερωμένος ε, τις επιλογές του και είναι μια βασική ελευθερία αυτή, την οποία εμείς υπερασπιζόμαστε. Γι' αυτό και υποβάλαμε τροπολογίες όσον αφορά την αναγνωσιμότητα και όπως είπα είναι ένα στοιχείο κλειδί γιατί μπορεί κανείς να έχει στην ετικέτα όλες τις πληροφορίες αλλά να μην μπορεί να τις διαβάσει. Έπειτα πρέπει να είναι πραγματικές, σωστές, να μην κοροϊδεύει κανείς τον καταναλωτή. Τι λιπαρά, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται σε ένα παγωτό ή σε ένα τυρί, αν είναι φυτικά ή όχι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κοροϊδεύσει κανείς τον καταναλωτή. Επίσης για τα προσυσκευασμένα. Πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές πληροφορίες για το φαγητό το οποίο ε, συσκευάζεται στο κατάστημα, εκεί μπορεί να υπάρχει εξαίρεση. Τώρα από τόσα ξέρουμε και ξέρουμε πολλά, ένα πράγμα που νοιάζει πολύ τον κόσμο είναι κυρίως το κρέας. Ο κόσμος τρομάζει, φοβάται για την υγεία του όσον αφορά το κρέας. Για τη δήλωση τώρα θρεπτικής αξίας επίσης. Εδώ έχω υποβάλει μία τροπολογία, γιατί εγώ νομίζω ότι ο κλάδος πρέπει να έχει μια κάποια ελευθερία τη στιγμή που οι συσκευασίε είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά σίγουρα ό,τι αναφέρεται συσκευασίε πρέπει να είναι κάτι απλό και να μπορεί εύκολα να το διαβάσει και να το καταλάβει ένας μεσαίος καταναλωτής. Το θέμα τώρα των αλκοολούχων ε, ποτών και των διάφορων ε, αναψυκτικών. Η άποψή μας είναι να μην δημιουργήσουμε υπερβολική γραφειοκρατία, ιδίως για τους μικρούς παραγωγούς. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια θέση που όλοι να έχουν να κερδίσουν από αυτήν όσο γίνεται περισσότερη προστασία για τον καταναλωτή δηλαδή από τη μια και από την άλλη να μην δημιουργούμε επιπλέον κόστος για την ε, βιομηχανία. Γιατί είμαι κατά του, των τριών χρωμάτων. Γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος άλλος να αποφασίζει για τον κόσμο τι θα τρώει. Να τους ενημερώνουμε, να τους δίνουμε πληροφορίες, να τους λέμε τι έχει μέσα, τι συστατικά περιλαμβάνει αυτό που αγοράζουν, αλλά μην είμαστε εμεί αυτοί που αποφασίζουν. Και το τι χρειάζεται ο δικό σα οργανισμό μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που χρειάζεται ο δικό μου ή τα παιδιά μα. Είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μα. Έχουμε διαφορετικέ ανάγκε και διαφορετικού τρόπου ζωή στο κάτω-κάτω. Και διαφορετικό προπολογισμό ο καθένα μα για τα τρόφιμα που αγοράζουμε. Οπότε όταν σε κάποιον βάλουμε ένα κόκκινο χρώμα, δεν είναι δικιά μα δουλειά αυτή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αφήνουμε την ελευθερία στους καταναλωτές Οπότε το θέμα αυτό του κόκκινο, κίτρινο, πράσινο δεν είναι τόσο αν συμφωνούμε, τι συμφωνούμε, όσο το τι άποψη έχει κανείς για τον καταναλωτή, αν πιστεύουμε ότι πρόκειται για έναν ελεύθερο και υπεύθυνο άνθρωπο. Εγώ θέλω να δώσω στον καταναλωτή όσο γίνεται περισσότερα μέσα για να μπορεί να κάνει μια σωστή για αυτόν επιλογή, αλλά να είναι αυτός που την κάνει την επιλογή και όχι εμείς ανταυτού. Για τα αλκοολούχα ποτά πάλι συμφωνώ για το ότι πρέπει να καλύπτονται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεικτά ποτά, ε, με αλκοόλ, τα αλκοπρόπς που λέμε, που τα χρησιμοποιούν πολλοί νέοι. Αλλά πρέπει να υπάρχει συνοχή στη στάση μας. Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις για τον ίνο, για το κρασί. Ένα μέρος καλύπτεται, ένα μέρος δεν καλύπτεται. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν. Να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να έχουμε σε πέντε χρόνια κάτι καινούριο, είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Δεν σημαίνει ότι δεν μας νοιάζει η υγεία των νέων. Σημαίνει ότι αυτός είναι ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε που είναι καλύτερος. Γιατί οι θρεπτικές αξίες σε ένα αλκοολούχο ποτό δεν είναι ίδια. Στο ουίσκι σε ένα κομμάτι φαγητό. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και να περιμένουμε. Κατά τα συμφωνώ με την Κρίστελ να παραμείνουμε σε μια γενική συζήτηση, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιο θέλει κάποια λεπτομέρεια για κάποια συγκεκριμένη τροπολογία, ευχαρίστω. Τώρα, όσον αφορά τι εθνικέ διατάξει, εμεί θέλουμε εδώ να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Οτιδήποτε κατακαιρματίζει την αγορά μα είναι κακό για τη βιομηχανία και για τον καταναλωτή. Οπότε ευχαρίστως να δούμε για το κεφάλαιο 6 και 7 τι θα κάνουμε. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερα από τα κεφάλαια 6 και 7. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Και συγγνώμη που στην αρχή δεν σας πρόσεχα, αλλά ναι, άκουγα τι μου έλεγε η γραμματεία. Και γιατί. Γιατί η γραμματεία μόλις μου είπε ότι έχουμε ένα νέο μέλος για πρώτη φορά εδώ που ήθελα να καλωσορίσω. Γι' αυτό το συζητούσα με τη γραμματεία. Για να προφέρω το όνομά σας σωστά. Η κυρία Μονιθακία από την Ισπανία που αντικαθιστά την κυρβαρία. Ελπίζω να πρόφερα κάπως σωστά το όνομά σας. Ο κύριος Κόσμος δεν είναι εδώ, δεν ξέρω αν θα έρθει. Και αν είναι κανείς άλλος από τους φιλελεύθερους εδώ. Τυρών όμως τώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Τυρών. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα και αργά, λέει ο μιλήτρια, για να μπορέσουν οι διερμηνείς να με μεταφράσουν καλά. Θα ήθελα καταρχήν θα ήθελα καταρχήν να επενέσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της και να πω ότι εμείς οι πράσινοι ε, σε πολλά σημεία συμφωνούμε με τις θέσεις ε, της εισηγήτριας. Νομίζουμε ότι πολύ σωστά ασχολείται με την ε, βάση της οδηγίας αυτής. Θέλουμε δηλαδή να επικαιροποιήσουμε τους ισχύοντες κανόνε για την ενημέρωση για τα τρόφιμα και θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει στους καταναλωτές ε, να κάνουν τις σωστές επιλογές στον αγώνα κατά των ε, ασθενειών που ε, συνδέονται με τον τρόπο ζωής. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες σχετικά με το ενόπνευμα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροπολογίες. Θέλουμε χρόνο να τις εξετάσουμε προσεκτικά. Ε, μία σημείωση, δεν είχαμε χρόνο να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες ε, προσεκτικά. Θα ήταν ε, πολύ πιο χρήσιμη η συζήτηση εάν είχαμε το χρόνο. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε συμβιβασμούς, αλλά όπως σας είπαμε το αλκοόλ έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά θα ήθελα να συζητήσω το βασικό θέμα, το, λεγόμενο σύστημα φανάρι, το, τους χρωματικούς κωδικούς σε σχέση με τις ε, πληροφορίες ε, διατροφικής αξίας. Τρία πράγματα θα πρέπει να εξετάσουμε. Τι λέει η επιστήμη, τι λένε οι οργανώσεις καταναλωτών και οι οργανώσεις υγείας και τρίτον, τι μας λένε οι εμπειρίες από τη ζωή. Το πρώτο, η επιστήμη. Δεν έχει γίνει πολλή δουλειά, αλλά έχουμε κάποιες έρευνες από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και διαπιστώνεται ότι για τους καταναλωτές είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε το σύστημα ε, φανάρι. έχουν γίνει δοκιμές με καταναλωτές. Ε, νομίζω ότι ε, είναι χρήσιμο να το έχουμε αυτό υπόψη μας κατά τις συζητήσεις μας. Δεύτερον, τι λένε οι οργανώσεις καταναλωτών, τι λένε οι οργανώσεις για την υγεία. Συμφωνούν απορρίπτουν το σύστημα διατροφικής αξίας, ε, λένε ότι είναι υπερβολικά τυποποιημένο. Τι είναι, ε, το, ε, ποιο είναι το μέγεθος μιας μερίδας και ποιος είναι ο μέσος άνθρωπος. Οι οργανώσεις κατανοτών της Ευρώπης, οι οργανώσεις καταπολέμησης του καρκίνου, το, της Ένωσης για τις καρδιακές παθήσεις, τέτοιες μη κυβερνητικές οργανώσεις μας λένε ότι για την υγεία των ανθρώπων είναι πιο χρήσιμο το σύστημα φανάρι, κόκκινο, και πράσινο, η χρωματική κωδική. Και όσον αφορά το σύστημα διατροφική αξία, να κοιτάξουμε τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δέκα χρόνια μπροστά από εμά βρίσκονται. Τώρα σιγά σιγά οι Ηνωμένε Πολιτείε εγκαταλείπουν το σύστημα διατροφικής αξίας και το, ε, έχουν στρέψει τα μάτια προς το Ηνωμένο Βασίλειο που στρέφεται προς ένα σύστημα χρωματικών κωδικών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε διαπιστώνουν ότι μετά από 10 χρόνια ότι αυτό το σύστημα δεν μας έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και άλλων ασθενειών που συνδέονται με τον τρόπο ζωής. Αυτό λοιπόν βρίσκω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισάγει ένα σύστημα το οποίο εγκαταλείπουν τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, θα είμαστε ε, ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε μαζί την επιστήμη, ε, της συστάσει διάφορων οργανώσεων και τις εμπειρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν καλοί τρόποι, να... δεν βλέπω να υπάρχουν καλοί λόγοι να εισάγουμε ένα τέτοιο σύστημα ευρωπαϊκό διατροφικής αξίας. Έχουμε λοιπόν υποβάλει τροπολογία σχετική. Και επίσης, δεν είμαστε τελείω ηλίθιοι, βλέπουμε τα σημάδια των καιρών, βλέπουμε ποιε είναι οι θέσει των ανθρώπων ε, στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Και να πω Τώρα που σας είπα σαφώς ποια είναι η θέση μας, είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε συμβιβασμούς. Δεν ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, ήρθαμε εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε αποτελέσματα στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ε, γι' αυτό στην συζήτηση ε, που θα έχουμε με τις κοιόδους εισηγητές ε, θα το έχουμε υπόψη μας αυτό. Απλά ήθελα να σας παρουσιάσω σαφώς τις θέσεις μας. Και επίσης, η Κρίστελ τώρα μόλις μου επισήμανε ότι υπάρχει και ένα τρίτο πρότυπο που πρότεινε ο κύριος Κρόιτσμαν τροπολογία υπαριθμών 282 που είναι η τρίτη λύση κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ε, σε ποια θέματα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πρόκειται λοιπόν για πρόσκληση και υποστήριξη της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πολύ σαφείς. Ε, εάν ε, μου το επιτρέπει η Επιτροπή, η Συγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές, ε, ε, μου επιτρέψουν να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Κλάρκιν, να σας μιλήσω για κάποιες από τις τροπολογίες που επεξεργάστηκε η σκιώδης εισηγήτρια της δικής μου ομάδας. Γενικά, στηρίζουμε τη θέση του ΕΛΚ σχετικά με το ότι τα αλκοολούχα αποτελούν ειδική περίπτωση και θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά για τα προϊόντα αυτά λόγω της ειδική τους φύσης. Όσον αφορά την ε, ευκρίνεια ε, της ε, συσκευασίας. Είμαι βέβαιος ότι εδώ υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, παρουσίαση των πληροφοριών ιδιαίτερα σε μικρές συσκευασίες, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητική η λύση που εφαρμόζεται. Θα πρέπει να γίνει συμβιβασμός ε, λαμβάνοντα υπόψη φοριών και τον χώρο που υπάρχει, διότι αλλιώς ε, θα παρουσιαστεί το πρόβλημα του υπερβολικού όγκου των πληροφοριών, κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το θέμα με το σύστημα φανάρι είναι μάλλον ότι υπεραπλουστεύει τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και εδώ συμβιβασμό. Θα ήθελα να ξέρω εάν είναι ένα θέμα που αφορά ειδικά τη χώρα μου, έχει να κάνει με την ευκρίνεια. Οι θερμίδες είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα μέτρησης της ενεργειακής αξίας. Θέλουμε λοιπόν ε, να είναι κατανοητό το σύστημα. Έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις που συνδέονται με την επισήμανση του κρέατος αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα του καταναλωτέ, όπω είπε και η κυρία Μπίλτ. Υπάρχουν αρκετέ περιπτώσει ε, τροφίμων, όπω για παράδειγμα τα προϊόντα ε, κοτόπουλου που μπορεί να περιέχουν ε, πρωτεΐνες ε, χοιρινού ή βοηού κρέατος. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για τα θέματα αυτά και επανέρχομαι και στο θέμα των αλλεργιογόνων, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι αλλεργικοί στα προϊόντα χοιρινού κρέατος. Εάν λοιπόν σε ένα προϊόν ε, από κοτόπουλο έχει προσθεθεί λίπος από χοιρινό, θα πρέπει ο καταναλωτής να το γνωρίζει αυτό. Υπάρχουν εδώ πολύπλοκοι τομείς. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ αναφέρθηκε στην υποχρεωτική επισήμανση του κρέατος και στους εναρμονισμένους κανόνες για τα αλλεργιογόνα. Είναι κάτι λοιπόν με το οποίο συμφωνούμε και θα συμμετάσχουμε στις σχετικές συζητήσεις. Ε, γενικά παρακολουθούμε στενά το θέμα Και ε, μπορώ να πω εκ μέρους της κυρίας ότι με πολύ ενδιαφέρον θα συμμετάσχει στις μελλοντικές συζητήσεις. Αυτά λοιπόν, λοιπόν από τη δική μας πλευρά. Βλέπω ότι ο κύριος Κρόιτσμαν ε, ήρθε. Θέλετε να πάρετε μια ανάσα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έχει ζητήσει το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο όταν ε, θα είστε έτοιμος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, παρακαλώ. Ο κύριος Ντεγιόν είναι και ο συζητητής μας. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εμείς έχουμε διάφορα που προσπαθούμε να προσθέσουμε με τις τροπολογίες μας. Το κεντρικό σημείο είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορά. Είτε πρόκειται για μεγάλη είτε για μικρή επιχείρηση, μεγάλης μικρής κλίμακας ή αν είναι ένα σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι ότι όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ακολουθήσουν τους ίδιους κανόνες. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει οι κανόνες που θα βάλουμε να είναι τέτοιοι, ώστε ακόμα και για ένα μικρό μαγαζί να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Δηλαδή να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσει για παράδειγμα για το μέγεθος των γραμματοσυρών. Για μένα όντως μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις για μη συσκευασμένα προϊόντα και επίσης εξαιρέσει και για το αλκοόλ, για τα πνευματόδη ποτά. Όσον αφορά αυτά τα μείγματα ποτών που χρησιμοποιούν πολύ οι νέοι και να έχουν την εντύπωση ότι είναι καλά, δεν κάνουν κανένα κακό. Το Βέβαια είναι πάντως ότι πρέπει να έχουμε κανόνες οι οποίοι να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν. Για τους μικρούς ανεξάρτητους, λοιπόν, είναι σημαντικό να μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες. Γι' αυτό και έχουμε φροντίσει για κάποιες τροπολογίες κι εμείς. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες για τη γνωμοδότηση αυτή, ώστε να προχωρήσει. Πάντως για μένα το βασικό είναι ο μικρός επιχειρηματίας, να μπορέσει και αυτός να επιζήσει με, αυτούς, με αυτές τις ρυθμίσεις. Να είναι τέτοιες οι ρυθμίσεις, σίγουρα ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι καλός, αλλά πρέπει να μπορεί να τεθεί και σε εφαρμογή. Εξού και οι τροπολογίες μας. Τώρα για άλλα θέματα, για το θέμα του σηματοδότη. Και εδώ νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί με τις ρυθμίσεις μας. Έχουμε μιλήσει με νόσες καταναλωτών, ακούσαμε απόψεις για αυτό το σηματοδότη, άλλοι το θέλουν, άλλοι όχι. Η ιδέα με το σύστημα του σηματοδότη είναι ότι όποιος βλέπει κόκκινο σκέφτεται «Α, κακό», ενώ δεν είναι πάντα έτσι. Γι' αυτό ίσως πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι άλλο. Σίγουρα είναι περίπλοκο. Πάντως ας προσπαθήσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να μην δίνει την εντύπωση το σύστημα του σηματοδότη ότι α, αυτό είναι σίγουρα κακό. Και δεν είναι η μόνη λύση, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Επίσης να είμαστε ελαστικοί, να δώσουμε περιθώριο στους μικρούς επιχειρηματίες να προετοιμαστούν. Οι ρυθμίσεις μας να είναι τέτοιες που να είναι ξεκάθαρες για τον καταναλωτή τι συστατικά έχει ένα προϊόν. Και εξάλλου μην ξεχνάμε πόσες πια πληροφορίες μπορεί να ε, πάρει ο καταναλωτής και εμένα μου έχει τύχει ένα πακέτο να το πάρω, να το κοιτάξω, να δω τι λέει. Λέει κάτι για, για θερμίδες. Πολύ ωραία. Θερμίδες, άμα κάποιο θέλει να δυνατήσει, όμως δεν πρέπει να κοιτάξει μόνο το θέμα των ε, θερμίδων, πρέπει να δει και το θέμα των λιπαρών και πολλά άλλα. Οπότε είναι περίπλοκο πάντα το θέμα αυτό των πληροφοριών για τα τρόφιμα. Τώρα πρέπει να είναι στον μπροστινό μέρο ή όχι τη συσκευασίε. Ίσως οι θερμίδες να είναι στο μπροστινό μέρος και οι υπόλοιπε πληροφορίες στο πίσω μέρος του προϊόντος. Αυτά και από εκεί και πέρα, άμα θέλετε, τις τροπολογίες μα να τις συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κρόιτσμαν, που είναι σκιώδης εισηγητής για την Άλντα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αναφέρθηκαν. Οι υπερβολικές πληροφορίες δεν είναι πληροφορίες πια, δεν είναι ενημέρωση. Το είπαν όλοι με όσους συνομιλήσαμε, γι' αυτό θα πρέπει οι πληροφορίες προς τους καταναλωτές να είναι ευανάγνωστες, δεν θα πρέπει όμως να είναι και υπερβολικός ο όγκος, διότι τότε δεν είναι καθόλου χρήσιμες. Αυτός είναι ο στόχος της πρότασής μας που υποβάλαμε όσον αφορά τα μη συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει τουλάχιστον ε, να ε, γίνεται ενημέρωση για τα αλλεργιογόνα. Τίποτα άλλο όμως δεν είναι απαραίτητο και σκεφτήκαμε επίσης ότι ε, τα 100 μιλιγκράμμ ή 100 μιλιλίτρ θα πρέπει να είναι η βάση για να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία. Βέβαια η παραγωγή τσίχλας ε, λένε ότι όταν μιλάμε για 100 μιλιγράμμι ή 100 μιλιλίτερ, τότε έχουμε ε, ήδη καλύψει την, την, ε, την κατανάλωση τσίχλας για ένα μήνα ολόκληρο. αλλά βασικά ο καταναλωτής όταν βλέπει το προϊόν στο ράφι θα πρέπει σύντομα να μπορεί να έχει στοιχεία σε συγκρίσιμη βάση. Και γι' αυτό προτείνουμε 100 γραμμάρια ή 100 μιλιλίτρ. Αυτό μπορεί να παρουσιάζεται και με ε, διαγράμματα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου το εξή. Όταν ε, θεσπίζουμε έναν κανόνα εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ε, θα πρέπει να μπορεί αυτός να αναιρεθεί σε εθνικό επίπεδο. Αν επιτρέψουμε υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις, τότε κατά τη γνώμη μας έχουμε δημιουργήσει διπλή γραφειοκρατία. Δηλαδή ο καταναλωτή θα πρέπει από τη μία να ξέρει τι θέλει η Ευρώπη και από την άλλη να γνωρίζει τι επιτρέπουν ε, τα κράτη-μέλη. Ε, με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ε, ε, πηγαίνουμε ενάντια στο νόημα της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν οι ευρωπαϊκοί κανόνες να είναι υποχρεωτικοί για τα κράτη-μέλη. Η βασική αρχή κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι οι απαραίτητες πληροφορίες να δίνονται, όχι υπερβολικές πληροφορίες. Ε, υπάρχει και το επιχείρημα του μεγέθους της συσκευασίας, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί για να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις. Και μία ακόμα μικρή παρατήρηση σχετικά με τις διατροφικές πληροφορίες. Ε, για παράδειγμα για κροκέτες πατάτας ε, οι, οι θερμίδες που δίνονται είναι πριν ε, παρασκευαστούν ή μετά διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στις θερμίδες της κροκέτας, της πατάτας του υλικού που υπάρχει στη συσκευασία δηλαδή και στην έτοιμη κροκέτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι γίνεται αν ετοιμάσει ε, το γεύμα μεγάλα ή με νερό. Θα τα αφήσω αυτό το θέμα της πατάτας, όχι την ε, πολύ αρέσει. Ευχαριστώ πολύ τους Σκιώδης. Έχω τέσσερα μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Να εξετάσω ποιος είναι στον κατάλογο και αν θέλει να συμμετάσχει κι άλλος. Κύριο Σφανόκ, Σβάμπ, κυρία Βάιλερ και Στάιλερ και ο Μότι. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Ο κ. Χουανόκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη εισηγήτρια για την γνωμοδότηση και που ευθύ εξ αρχή είχε μέρημνα την προστασία και την ενημέρωση του καταναλωτού. Μας προτείνει πολλές ε, βελτιώσεις στο αρχικό κείμενο και ελπίζω να την υποστηρίξουν πολύ στην Επιτροπή διότι πρόκειται περί θέματος που αφορά την υγεία των πολιτών των Ευρωπαίων και πιο συγκεκριμένα εκείνων που δεν ενημερώνονται πάρα πολύ καλά, αυτοί που δεν, δεν γνωρίζουν τόσο καλά το θέμα. Έχω ένα ερωτηματικό που συμμερίζονται κι άλλοι. Η πρόταση χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα σηματοδότησης για την ενεργειακή περιεκτικότητα των τροφίμων αν τέτοιο χρωματικό κώδικα θέλουμε να είναι αποτελεσματικό όσον αφορά τον καταναλωτή που ήδη είναι ενήμερο, σε κάποιε χώρε η προστασία και ενημέρωση του καταναλωτού είναι λιγότερο ανεπτυγμένη και που οι καταναλωτέ εν γέννη είναι λιγότερο ενήμεροι, αυτό το σύστημα είναι υπεραπλουστευμένο και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Θα μπορούσε να οδηγήσει τον καταναλωτή να σταματήσει την κατανάλωση όλων των τροφίμων που έχουν κόκκινο σήμα, ενώ στι περιπτώσεις μια λογική κατανάλωση των λόγω προϊόντων δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα όσον αφορά την υγεία. Αντίστροφα θα μπορούσε να ευνοήσει την κατανάλωση τροφίμων που ε, είναι αμφισβητήσιμη η θετική του επίδραση στην υγεία. Ας πούμε θα μπορούσαν κάποια τρόφιμα να πάρουν πράσινο φως λόγω χαμηλή περιεκτικότητας σε θερμίδες ας πούμε ας πούμε η Coca-Cola Diet η οποία μέσα έχει ασπαρτάμι ε, αντί για ζάχαρη και μπορεί να ευνοεί την κατανάλωση αυτής. Λοιπόν, θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται η ενεργική περιεκτικότητα ε, η ενεργεια, το ενεργειακό περιεχόμενο των διαφόρων τροφίμων χωρίς να τα στιγματίζουμε. Για 100 γραμμάρια λοιπόν ή 100 μιλιλίτρα είναι η μόνη υποχρεωτική αναφορά και ίσως να μην είναι σχετική για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν τρόφιμα βάρους και όγκου που ποικίλει κατά πολύ. Προτείνω λοιπόν η ενεργειακή ε, τιμή να αναφέρεται συστηματικά κατά μερίδα ή στην περίπτωση ενός τροφίμου που δεν μπορεί να προσμετρηθεί με μερίδα σε βάση το καθαρό βάρος του προϊόντος έτσι ο καταναλωτής θα μπορεί να έχει πληροφορίες ακριβέστερες και πιο ευανάγνωστες και πιο εύληπτες. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σβάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η εντύπωση μου που επιβεβαιώθηκε μετά την τελευταία παρέμβαση είναι ότι η συζήτηση σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζω την ίδια συζήτηση από το παλιό κοινοβούλιο, από την παλιά θητεία και βλέπουμε όλο και πιο ε, πολύ την ε, θέση ότι δεν έχουμε μόνο τις ε, τους τρεις παράγοντες που ανέφερε η κυρία Τούρινεν, ναι, ναι, έχουμε και την κοινή λογική, η οποία μας λέει ότι τα αποτελέσματα, τον, οι εμπειρίε των Ηνωμένων Πολιτειών Δείχνουν ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί με βέλτιστο τρόπο. Αλλά το να βγάλει κατευθείαν το συμπέρασμα κανεί ότι το σύστημα φανάρι είναι καλύτερο, αυτό βρίσκω μάλλον ότι είναι αμφίβολο. Σε πολλές οριακές περιπτώσεις έχουμε δει ότι φτάνουμε στα όρια με το σύστημα που εφαρμόζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να είναι φιλικό προς τον καταναλωτή. Να αναφέρω ένα θέμα το οποίο ήδη θύχθηκε. Εγώ έρχομαι, προέρχομαι από το, από το μέλλον αδρυμό. Έχουμε εδώ ένα ειδικό ζαμπόν, το οποίο, του οποίου προστατεύεται η προέλευση. Ε, αλλά οι πρώτες ύλες προέρχονται από την ε, Ανατολική Γερμανία ή από άλλες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν ε, να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να προστατεύει την ε, ονομασία προέλευσης ε, του κρέατος, αλλά κάποιοι είπαν ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ορίσουμε τα κριτήρια για να γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω τι προτάσεις θα λάβουμε για να έχουμε ένα διαφανές σύστημα επισήμασης. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Σβάμπ. Η κυρία Βάιλερ. Äh, ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, δεν, θα έπαιρνα το λόγο ε, για το ενδιαφέρον αυτό θέμα της κυρίας Σάλτεμος, αν ε, η πρώτη παρέμβαση θα ήταν αυτή της κυρίας Σέμπιλτ. Εγώ δεν βρίσκω πολύ καλό να ε, μιλάμε τόσο επιθετικά για το σύστημα φανάρι. Βρίσκω ότι το σύστημα φανάρι είναι ένα πολύ καλό σύστημα, όχι σε όλους τους τομείς, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να το εξελίξουμε περαιτέρω. Εάν όμως πράγματι θέλουμε να ακούσουμε τους πολίτες και όχι μόνο τους Γερμανούς καταναλωτές, και, όχι μόνο οι Γερμανοί καταναλωτές θα θέλουν το σύστημα αυτό, οι Βρετανοί είναι ικανοποιημένοι με το θέμα αυτό και νομίζω ότι και ε, άλλα κράτη-μέλη θα ε, ε, ενδιαφέρονται. Εάν λοιπόν ακούμε τους πολίτες θα διαπιστώσουμε ότι θέλουν το σύστημα φανάρι. Ε, παρακαλώ λοιπόν να μην μιλάτε με τόσο επιθετικά λόγια ότι το σύστημα φανάρι είναι δικτατορικό. Και θα ήθελα και εδώ στον γείτονά μου προ τα αριστερά να πω ότι ναι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την κοινή λογική. Κάθε άνθρωπο, κάθε καταναλωτή, κάθε καταναλώτρια γνωρίζει πόση ζάχαρη υπάρχει στην Coca-Cola και πόσο λίπος υπάρχει στα chips ή στις τηγανιτές πατάτες. Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται ειδική ετικέτα. Ε, ως προς την ερώτηση τη Κρίστελ ε, Σάλτεμόζα σχετικά με ε, την γραφή Μπράι, ε, βρίσκω πολύ ωραία την ιδέα αυτή. Έχω έναν τυφλό μαθητή στην ε, δική μου εκλογική περιφέρεια, αλλά ε, είναι μεγάλος, μεγάλο το άχθος για τις επιχειρήσεις, ενδεχομένως να το εισάγουμε αυτό προαιρετικά. Η παραγωγή τροφίμων που θέλουν και μπορούν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό, μπορούν να το προσπαθήσουν σε προαιρετική βάση. Αυτό ίσως ε, να μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη λύση και άλλο πρόβλημα τα περιφερειακά προϊόντα. Όπως ε, όλοι σας, και στην πατρίδα μου έχουμε ε, προϊόντα της περιφέρειας τα οποία προωθούμε και θέλουμε οι καταναλωτές και για λόγους ε, περιβαλλοντικούς, λόγω των μεταφορών κλπ. θέλουμε να προτιμούν οι καταναλωτές τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα κρέας, λαχανικά, ε, φρούτα, ε, στα φρούτα ε, υπάρχουν οι ρυθμίσει αυτές. Δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο το κρατήδιο, θα πρέπει να αναφέρεται η περιοχή από την οποία προέρχονται, Καλαβρία, Νότια Ιταλία κλπ. κύριε Σφάπ, εγώ δεν είμαι τόσο μεγαλοψυχή όσο εσείς να λέω ότι ότι ε, έρχεται από την βόρεια έση το κρέας ε, από τον Μέλλον Αναδρυμό εάν το κρέας αυτό ε, ουσιαστικά προέρχεται από την Πολωνία ή από την, τη, τη στην Ανατολική Γερμανία, την Φραγκούρτη στον Όντερ. θα πρέπει Λοιπόν, να λάβουμε υπόψη μας και το επιχείρημα αυτό όσον αφορά την αγορά. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ε, να έχει παραχθεί στην ε, Ουγγαρία ή στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάλ. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Κρίσταλ για τη σκληρή δουλειά που έκανες. 280 τροπολογίες σου δόθηκαν την Παρασκευή και έκανε φοβερή δουλειά για να μα προτείνει αυτά που πρότεινε ε, μέχρι τώρα και ελπίζουμε στο μέλλον να σου δοθούν πιο γρήγορα τροπολογίε. Η κυρία Σβάιλερ αναφέρθηκε στα ε, προϊόντα των ε, εκμεταλλεύσεων με αναγραφή σε γλώσσα μπράι. Ίσως θα πρέπει να δούμε και την οδηγία για τους αγρότες. Εκεί είχαν ειδηθεί τροπολογίες για την μπράι. Και αν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε κάτι απλά, ίσως θα πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει προηγουμένως τι υπήρξε επιτυχές. Όσον αφορά τη χώρα προέλευσης, υποστηρίζω αυτά που υπόθηκαν. Είναι σημαντικό να εξεταστεί για το σύστημα αυτό της σηματοδότησης. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέποντας τι γίνεται όσον αφορά τις οργανώσεις καταναλωτών και προστασία της υγείας, όσον αφορά το σύστημα, φαίνεται ότι είναι το ευκολότερο και δημοφιλέστερο σύστημα που βοηθά τους καταναλωτές και δεν επιβάλλει τίποτα σε κανέναν. Αντίθετα, δίνει την ελευθερία στους καταναλωτές ενήμεροι να κάνουν την επιλογή τους και εγώ θεωρώ ότι αυτός ήταν ο στόχος της προτάσεως και αυτό που είναι ενδιαφέρον και δεν αναφέρθηκε στην Επιτροπή μας είναι και το εξή. Πολλές εταιρείε υιοθετούν το σύστημα αυτό της σηματοδότησης του φαναριού γιατί θεωρούν ότι είναι εμπορικά θετικό διότι θέλουν οι καταναλωτές να επιδιώξουν την υγεία, να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση με την γύρανση του πληθυσμού και όλα αυτά. Το θέλουν. Και πολλά από αυτά που κάνουμε σε αυτή την πρόταση αφορά τα προσυσκευασμένα προϊόντα, που στη δική μου εκλογική περιφέρεια τουλάχιστον αυτά τα αγοράζουν οι φτωχότεροι καταναλωτές. Και αν αυτοί που τα παράγουν, αν πιέσουμε αυτούς που παράγουν τα προϊόντα να τα κάνουν υγιέστερα, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα όπως είναι καρδιακά ε, προβλήματα για τις δόσεις είναι ντροπή ότι αυτοί που παράγουν δημητριακά δεν ασχολούνται σωστά με το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα έξοχο έγγραφο με τίτλο «Ε, «Αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο στον τομέα των δημητριακών». Όσον αφορά τις δόσεις, τις ε, μερίδες πρέπει να γίνει κάτι. Όσον αφορά το αλκοόλ, δεν θα μπορούμε να ζητήσουμε από τους Σκοτσέζους ε, να βάλουν ετικετοθεσία όσον αφορά τα μιλίτρα στο whisky. Δεν θα πρέπει όμω να τη γλιτώσουν οι παραγωγοί νοπνευματοδών εντελώ. Την περασμένη εβδομάδα στη Σκωτία αναφέρθηκαν τα αλκοολικά ποτά που έχουν μέσα καφέινη. Στο Strathclyde η αστυνομία έδειξε ότι σε 100.000 περιπτώσει τα καφεϊνούχα αλκοολικά ποτά δεν αναφέρουν, όπω είναι το Bockfast που αναφέρατε. Αυτά τα ποτά επηρεάζουν τι κοινότητέ μα, οδηγούν σε αντικοινωνική συμπεριφορά αυτά τα αλκοούχα ποτά με καφέινη πρέπει τα πιο ακαθόδη προϊόντα να τα αντιμετωπίσουμε. Και ίσως υπάρχει η ευκαιρία τώρα να το κάνουμε αυτό, να ζητήσουμε απαγόρευση, κάποιοι ζητούν απαγόρευση των καφεϊνούχων αλκοολικών ποτών. Αυτό ζητούν στη δική μου εκλογική περιφέρεια, ίσως και άλλοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Η Κρίσταλ μπορεί να μας πει τι γίνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι ξέρω αυτή είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση, είναι πάρα πολύ σημαντικά, άμεσα με πολλά θέματα που αφορούν τους ε, πολίτες μας και ελπίζω ότι τους επόμενους, επόμενες εβδομάδες και μήνες θα λύσουμε τις διαφορές μας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο ο κύριος Μότι. Κύριε Κρότσφελτ, κύριε Κοράτσα θέλετε να μιλήσετε τώρα. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, αν θέλω να πάρω το λόγο. Ο κύριος Μότι, πρώτα. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο, συμμετέχω στη συζήτηση που αφορά το χρωματικό κώδικα, όπως ακαλείται, αυτό το σηματοδότη. Διότι πιστεύω ότι επειδή η δική μας Επιτροπή ασχολείται με την υπεράσπιση των καταναλωτών, όλοι έχουμε κοινό στόχο και καμιά φορά ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα φαίνεται ότι διαφέρει, αλλά θα πρέπει να αναλυθεί για να δούμε ποιος είναι ο τελικός σκοπός. Όλοι στη, θέλουμε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν μια επιλογή που βασίζεται στη γνώση και σε συγκεκριμένα κριτήρια. Όταν ακούω να λέμε ότι κάποιες εταιρείε διάλεξαν ένα χρωματικό κώδικα διότι θεωρούν ότι αυτό οδηγεί σε εμπορικό πλεονέκτημα, το πιστεύω. Διότι επιλεγεί και διαλέγει μία παράμετρο που αναφέρει, α πούμε, θερμιδική περιεχόμενο σε θερμίδε, αν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε να προξενήσουμε σύγχυση. Διότι άκουσα πολλέ φορέ να αναφερόμαστε σε υγιεινή διατροφή και να εντοπίζουμε τι θερμίδε, να ταυτίζονται οι θερμίδε τελικά, υψηλή μπορεί να συνδέσουμε μεγάλη περιεκτικότητα σε θερμίδες σαν ε, ανθυγιεινή διατροφή και λίγες θερμίδες σαν υγιεινή. Δεν ισχύουν αυτό. Είδαμε στη ΣΥΠΑ, έγιναν κάποιες έρευνες ε, που δείχνουν ότι είναι τα αποτελέσματα. Στη ΣΥΠΑ απομακρύνονται από την ετικέτα με τις, με δοσολογίες ε, που προτείνονται. Και γιατί γίνεται αυτό πρέπει να δούμε. Ίσως να είναι εσφαλμένη προσέγγιση ε, διότι, να πούμε, διότι υπάρχουν πολλοί παχύσαρκοι και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι να δούμε πώς κάνουν οι Αμερικανοί την επιλογή τους βάσει ποιων κριτηρίων, σε ποιο πλαίσιο ε, κοινωνικό, πολιτισμικό. Διαφορετικά η ετικετά θα γίνει ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Θα δίνει άπειρη σειρά πληροφοριών, πολύ χρήσιμες πληροφορίες μένουν για τους καταναλωτές θα είναι, αλλά πού να μπουν σε μια ετικέτα τους πληροφορίες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν άλλα μέσα και άλλα συστήματα. Ας πούμε, ε, το μαϊντανό σε μεγάλες ποσότητες ε, μπορεί, κάνει κακό στο σηκώτη. Εάν ε, ένα παιδί μικρό φάει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, πιθανότητα θα πεθάνει. Αυτή είναι πληροφορία που ε, είναι πολιτισμική προσέγγιση όσον αφορά την ε, κατανάλωση. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στις μητέρες ότι δεν μπορούν να κάνουν ένα παιδί να φάει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες του μετανού. Νομίζω ότι η ιδέα που θα πρέπει να είναι στη βάση των εργασιών μας θα πρέπει να είναι να δώσουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό πληροφοριών που μπορούν να μπουν σε μια ετικέτα χωρίς να αντικαταστήσουμε καταστήσουμε όμως τη δυνατότητα επιλογής του καταναλωτού που θα πρέπει να κάνει επιλογή λαμβάνοντα σειρά άλλων πληροφοριών που μπορεί να μαζέψει από άλλου φορεί όπω είναι ε, οι ενώσει προστασία καταναλωτών. Πληροφορίε που μπορεί να διαθέσω στον καταναλωτή. Ένα άλλο παράδειγμα. Καμιά φορά με την υπερβολή καταλαβαίνουμε το παράδειγμα. Μιλήσαμε για χρώματα, χρωματικό κώδικα, αλλά και γραφικά. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον κωδικό αυτό του σηματοδότη με ένα γραφικό χαρακτήρα ε, σήμα που θα βάζει νεκροκεφαλή, παραδείγματο χάρη, άμα έχει πολλέ θερμίδε. Σύμβολο του θανάτου. Να πούμε στον καταναλωτή, κοιτάξτε, αυτό το στοιχείο το θερμιδικό μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό. Όπω το κόκκινο σηματοδότη, όταν βλέπουμε κόκκινο φω στο σηματοδότη, σταματάμε. Πήγα στην υπερβολή να σα δείξω ποια είναι η έννοια. Με ένα σηματοδότη λέμε σταμάτα. Αλλά δεν εκφράζουμε απαραίτητα μία κρίση όσον αφορά το προϊόν αν είναι υγιές ή όχι. Λέμε ότι αυτό το προϊόν λίγο πολύ ε, έχει πολλές θερμίδες. Αν τώρα ένα παραγωγός, όπως ξεκίνησα κλείνω, αν ήμουν παραγωγός θα ήθελα να έχω το χρωματικό κώδικα εάν παρήγαγα ένα ανθρακούχο ποτό που δεν είναι πολύ υγιεινό αλλά με περιεχόμενο τεχνητή, τεχνητής ουσία και όχι ζάχαρη, διότι θα παίρναγε με πράσινο φως γιατί δεν έχει πολύ ζάχαρη και θα, να το παρουσιάσουμε αυτό και να μιλάμε στου καταναλωτέ για υγιεινή διατροφή είναι διαφορετική προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ ανεκτικό διότι χάσαμε ένα σημείο, άρα έχουμε παραπάνω χρόνο. Κυρία Βανιού, η Αντιπρόεδρος τι θα συμβάλλει. Η κυρία Κοράτσα Φέλτ ε, θέλετε να παρέμβετε για δεύτερη φορά. Ας ξεκινήσουμε από την κυρία Βανιού και μετά την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δώσω στη σκιώδη συγγήτρια την δυνατότητα να συνοψίσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να αφήσω χρόνο για την εισηγήτρια την οποία και συγχαίρω και θαυμάζω το κουράγιο της γιατί με τόσες πολλές τροπολογίες που πάνε προς πάσα κατεύθυνση, όπως είπαμε δεν είναι εύκολο. Μπράβο της λοιπόν. Πρέπει να συμφωνήσουμε τι προσπαθούμε να πετύχουμε όλοι μαζί. Οι καταναλωτές, οι πολίτες πρέπει να έχουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες στη διάθεσή τους. Από εκεί και πέρα μπορούμε και να δουλέψουμε πάνω στην οτροπία της επόμενης γενιάς να καταναλώνει λιγότερο, να καταναλώνει με περισσότερο ευφύ τρόπο. Εγώ το έχω σκεφτεί πολύ αυτό το θέμα του σηματοδότη. Στην αρχή ήμουν πολύ υπέρ, μετά όμως σκέφτηκα όχι, είναι πολύ περιοριστικό αυτό το σύστημα του σηματοδότη. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο, ώστε σε κάθε προϊόν να έχουμε τα βασικά, δηλαδή λιπαρά, ε, ζάχαρη, αλλεργιογόνα εννοείται, αναμερίδα ή ανα 100 γραμμάρια, έτσι ώστε ο καθένας μας να μπορεί να έχει την εικόνα του τι αγοράζει. Και μετά να πει, α, αν αγοράζω αυτό, εντάξει, αλλά επειδή είναι λιπαρός, αγοράσω κάτι άλλο που είναι λιγότερο λιπαρός ή χρόνος. Πρέπει να έχουμε τα βασικά στοιχεία με τα χρώματα, εντάξει, να βάλουμε ένα χρώμα για τα λιπαρά, ένα για τη ζάχαρη, αλλά όχι απαραίτητα αυτό το κόκκινο, κίτρινο, πράσινο που το κόκκινο σημαίνει απαγορεύεται. Γιατί τότε θα πρέπει να τα βάλουμε και στην Coca-Cola Light. Γιατί όντω λέμε δεν έχει μεν ζάχαρη, ναι, αλλά έχει ασπαρτάμι που είναι επικίνδυνη. Οπότε δεν νομίζω ότι εμεί μπορούμε να επιτρέψουμε στου εαυτού μα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαγορεύσουμε το ένα ή το άλλο προϊόν ή αντίθετα να πούμε ναι, πράσινο φω για το ένα ή το άλλο προϊόν. Όχι, νομίζω ότι ο κάθε καταναλωτή πρέπει να γνωρίζει τι αγοράζει, αυτό αν ναι, και όντα ενημερωμένο να καταναλώνει βάσει της επιλογής του για να προστατεύσει όπως πιστεύει καλύτερα την υγεία του. Παρακαλώ, η κυρία Κορατσαμπίλτ. Εντάξει, νομίζω ότι ο κύριο Μότι και άλλοι με κάλυψαν λίγο πολύ. Πάντω, θέλω να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα Βίλερ που μου έδωσε την ευκαιρία να εξηγήσω λίγο καλύτερα ναι, όντω, όντω είμαι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είμαι επιθετική, αλλά όντω έχω στην καρδιά μου αυτό το θέμα. Για τα 9 χρόνια τη ζωή μου έχω περάσει κυρίω στη Σουηδία, στι βόρειε χώρε πάντω γενικότερα, για να μιλάω για τα τρόφιμα και τη διατροφή και να προσπαθήσω να προωθήσω τα τρόφιμα ποιότητα με σεμινάρια, στα σούπερ μάρκετ και αλλού. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ε, μιλάνε εκ μέρου των καταναλωτών και λένε ότι είναι υπέρ του συστήματος του σηματοδότη, δεν είναι η εμπειρία που έχω εγώ. Γιατί ο καταναλωτής φυσικά και θέλει κάτι όσο γίνεται πιο απλό και θέλει να ανακουφίζεται, να μην έχει βαριά δουλειά να κάνει όταν ψωνίζει. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε κάτι περιορισμένο. Όταν ο καταναλωτής έχει την πραγματική ενημέρωση και αν του δίνουμε κάτι υπερβολικά επιφανειακό, δεν του αρέσει γιατί δεν έχει αρκετέ πληροφορίε. Ορισμένοι μπορεί να προτιμάνε σήμερα και να λένε ότι προτιμά το σύστημα του σηματοδότη επειδή δεν έχουν τι πληροφορίε που θα θέλανε. Αν όμω του δώσουμε τι πληροφορίε που θέλουν, θα νιώσουν εμπιστοσύνη σε αυτέ και του φτάνουν. Όλοι θέλουμε να δώσουμε στα χέρια του καταναλωτή κάποια δύναμη και να τον βοηθήσουμε να αποφασίζει για την υγεία του. Δεν μπορούμε να πούμε εμεί από μόνοι μα ότι η ζάχαρη, τα λιπαρά, έξω ότι είναι κακά για την υγεία. Εξαρτάται από την ποσότητα, εξαρτάται από το ποιο τα καταναλώνει. Γι' αυτό εγώ επιμένω. Σοκολάτα για παράδειγμα. Εγώ τρώω πολύ γιατί μου κάνει καλό. Μου δίνει ενέργεια, με βοηθάει. Και είναι πολύ υγιεινό για μένα. Έχει μαγνήσιο, έχει κανεί αντίρρηση. Νόστιμο βεβαίω. Λοιπόν, Ό,τι και να μου πείτε εσείς, εγώ σοκολάτα θα τρώω. Και θα δίνω και βούτυρο στα παιδιά μου. Γιατί το βούτυρο είναι καλό για τα παιδιά. Έχει πολλές βιταμίνες. Α, για παράδειγμα. Εγώ μεγάλωσα ε, ακούγοντα τον πατέρα μου να μου λέει μη βγάζετε το λίπος από το ζαμπόν πάρμα. Όχι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας δώσω, οπότε επιμένω και θα συνεχίσω τον αγώνα μου κατά του συστήματος του σηματοδότη. Πρόεδρος, σας επέτρεψα να δευτερολογήσετε και η κυρία Τούριν όμω θέλει επίσης να πάρει και πάλι το λόγο. Ναι, είσαστε όμως παρακαλώ σύντομοι. Ναι, ναι, θα είμαι. Είναι πολύ επικίνδυνο να γενικεύουμε ο καθένας την προσωπική του εμπειρία και να την παρουσιάζει εδώ σαν ένα εμπειρία ολόκληρης της κοινωνίας. Εντάξει, Μπορείτε εσείς να βασιστείτε στη δικιά σας εμπειρία και καλά κάνετε. Και εγώ το κάνω. Τη δικιά μου την εμπειρία τη χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου. Αλλά πρέπει από εκεί και πέρα να τη συνδυάσουμε και με τους υπόλοιπους. Και εκεί είναι που πάει στραβά το πράγμα. Δεν το κάνετε. Θα ήθελα εσείς να μου δείξετε το ΕΛΚ για τη δουλειά που θα κάνουμε στη συνέχεια. Γιατί πρέπει να συστήσουμε το δικό σας το σύστημα. Εγώ ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω, δεν το βλέπω. Εγώ δεν λέω ότι επιμένω υπέρ κατά του σηματοδότη, γιατί έτσι κι δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν ένα σωρό άλλε πτυχέ, ε, νοοτροπία κλπ. Συμφωνώ απόλυτα. Όμω, α δούμε τα γεγονότα καταρχήν και από τα γεγονότα καταλήξουμε σε επιλογές βασιζόμενοι και στην εμπειρία αλλά και στην επιστήμη να δούμε τι έχουν κάνει άλλε χώρες για να λύσουν αυτό το ζήτημα. Και εγώ θα συνεχίσω να τρώω σοκολάτα πάντως, να ξέρετε. Δεν θα τη σταματήσω. Ωραία, λέει ο πρόεδρο. Πολύ χαίρομαι που σας αρέσει η σοκολάτα. Έχω μια εταιρεία στη δικά μου εκλογική μου περιφέρεια, πολύ κοντά εκεί που μένω και ακούμε μάλιστα πολλέ εφημερίδες τελευταία από εκεί Χαίρομαι λοιπόν που σας αρέσει η σοκολάτα. Πάντως, εγώ αυτό που ακούω και μου λένε και οι γιατροί ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός και όντως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι λέμε. Γιατί μπορεί να μας αρέσει ολονών να τρώμε λίγη σοκολάτα, αλλά δεν ζούμε από τη σοκολάτα. Συγγνώμη που δεν έχω καλωσορίσει εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μαθιουδάκης είναι που θα πάρει το λόγο, έτσι δεν είναι. Και καλωσορίζω εδώ και το Συμβούλιο, κυρίως τον κύριο Κάρλος Κρέσπο που ήρθε, εκ μέρου της Ισπανική Προεδρία. Αν και αυτό θέλει το λόγο μετά, ευχαρίστω. Αλλά ίσω να μην θέλει. Πρώτα όμω, ο κύριος Μαθιουδάκης. Παρακαλώ. Πείτε μας τη γνώμη σα για τόσα ακούσατε εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Την άκουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την μέγιστη προσοχή. Ο τόνος δόθηκε από τις αρχικές παρατηρήσεις της εισηγήτριας της κυρίας Αλτεμός που είπε ότι είναι δύσκολο να πει κανείς οτιδήποτε σχετικά με την κατεύθυνση που θα λάβουν διάφορα ζητήματα λόγω απόκλησης απόψεων. Απ' την άλλη, εντυπωσιαστήκαμε από την πολιτική συμφωνία περί του σκοπού της ε, προτάσεως. Δηλαδή, να προστατευθούν οι καταναλωτές, να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέξουν και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε με όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να διαμορφωθεί σε επόμενες μέρες. Να έχουμε νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε λίγες μέρες. Και είναι δύσκολο λόγω της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα σχετικά με τα υποθέντα. Ακούσατε τα όσα είπε ο ψήφιος ε, Επίτροπος Ντάλι στην Ακρόαση. Δύο ήταν τα σημαντικά που πρέπει να συγκρατήσουμε. Πρώτον, ότι τα συμφέροντα του καταναλωτού θα έχουν ύψιστη προτεραιότητα για αυτόν. Και δεύτερον, ότι προτίθεται να ενημερώσει τους καταναλωτές να γνωρίζουν τι τρώνε αλλά να μην τους λέει τι να φάνε. Νομίζω λοιπόν ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαμορφωθεί από αυτά που δηλώθηκαν. Κάτι άλλο που συγκρατούμε από τη σημερινή συζήτηση. Είναι το σχόλιο της κυρίας Κοράτσα. Είπε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ενοπνευματόδη είναι λογική. Την ευχαριστούμε για το σχόλιο. Πιστεύουμε όμως ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι προτάσεις μας είναι λογικές και σε πολλούς άλλους τομείς από αυτούς που συζητήθηκαν. Μπορώ να αναφέρω κάποια σημεία. Αναφέρθηκε η χρωματική σηματοδότηση εκτενώς. Υπάρχει πρότασή μας σχετική και είναι λογική προσέγγιση διότι αναγνωρίζεται αυτό που ανέφερε ο κ. Ντεγιόγκ. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Και αυτό που είναι λογικό και αποδεκτό σήμερα από κάποιους καταναλωτές, ίσως να μην είναι για όλους τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η πρότασή μας όσον αφορά την παρουσίαση των πληροφοριών για το διατροφικό περιεχόμενο είναι κάτι που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους ε, μπλεκομένους φορείς και με την συμβολή των αρμοδίων αρχών. Αυτό θα ήταν λογικό, διότι θα επέτρεπε να κάνουμε δοκιμές όσον αφορά αυτές τις μεθόδους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην ευρωπαϊκή αγορά και στους ευρωπαίους καταναλωτές και έτσι ίσως να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό τρόπο παρουσίασης. Έγινε συγκεκριμένη η πρόταση για το πώς θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες, το σύστημα GDA και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές και να έχουν επιλογή. Δεν λέω ότι θα καταλαβαίνουν όλοι οι καταναλωτές όλες τις πληροφορίες. Αναφέρθηκε όμως και η εκπαίδευση που θα πρέπει να συνοδεύει τους ε, κανόνες που θα υιοθετήσουμε. Ενημέρωση δηλαδή. Συζητήθηκε και το θέμα της χώρας προέλευσης και η κυρία Κοράτσα είπε κάτι που είναι σημαντικό. Είπε ότι ο κόσμος θέλει να ξέρει από πού προέρχεται το κρέας. Διότι ο κόσμος φοβάται για την υγεία του. Το Κοινοβούλιο, παρακαλώ, ας το εξετάσει, ας διώξει αυτή την ιδέα ότι η ετικέτα της χώρας προέλευσης συνδέεται με θέματα υγείας. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια. Κριτήρια που εξασφαλίζουν το ότι είναι ασφαλή προς κατανάλωση. Και η ετικετοθεσία που αφορά τη χώρα προέλευσης δεν πρέπει να διασυνδέεται με πτυχές υγείας ή πτυχές μικροβιολογικές σχετικά με το προϊόν. Πιστεύουμε και πάλι ότι η πρότασή μας είναι λογική. Διότι προτιθέμεθα να δώσουμε τις πληροφορίες αυτές στον καταναλώτη όταν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ούτως ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και οι πληροφορίες πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Όσον αφορά την εθνική νομοθεσία που ανέφεραν πολλοί από εσά ότι θα πρέπει να παραμείνει να σημειώσω ότι έχουμε ήδη κανόνες που υφίστανται. Δεν εισάγουμε κάτι νέο. Ίσως το Συμβούλιο να έχει να πει κάτι σχετικά με το ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εδώ μπορώ να σταματήσω. Δεν θα ήθελα να επισέθω σε λεπτομέρειες επί κάθε σημείου, διότι δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαθιουδάκη. Νομίζω ότι ήταν πολύ λογική η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πάντα το Κοινοβούλιο μπορεί να βελτιώνει τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δίκαιο να το πούμε αυτό. Ο κύριο Κρέσπο δεν θέλει να πάρει το λόγο. Θέλετε, θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και έχω την τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα μου που έχει αναλάβει την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες μας όσον αφορά την υπόθεση αυτή τον Ιανουάριο σε μια δίμερη συνεδρίαση και έχουμε προγραμματίσει και νέες συνεδριάσεις για το εξάμεινο αυτό. Έχουμε εξετάσει το θέμα των ετικετών στα προϊόντα. Θα συνεχίσουμε βάσει του κειμένου που μας είχε αφήσει η Σουηδική Προεδρία και την οποία ευχαριστώ για τις προσπάθειές της. Όσον αφορά τους στόχους τώρα της δικιάς μας Προεδρίας δεν θέλω να επεκταθώ. Έτσι κι αλλιώς θα έρθει εδώ ο Υπουργός μεθαύριο, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί του γι' αυτά. Το μόνο που θέλω είναι να πω στους συζητητές και τους κοιόδης ότι είμαι στην διάθεσή τους για οποιαδήποτε συζήτηση θέλουν να έχουμε μαζί και ότι ανταλλαγή απόψεων θέλουν, ευχαρίστω. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρέσπο και εσά και του συναδέλφου σα από το Συμβούλιο που ήρθατε εδώ σήμερα. Τώρα η κυρία Σαλτεμόζα θα έχει το λόγο και πάλι για να ολοκληρώσουμε όσον αφορά αυτό το σημείο και να συζητήσουμε λίγο ίσω και τι προθεσμίε, ε? και ό,τι άλλο διοικητικό υπάρχει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνοψίσω. Σήμερα δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να συνοψίσω τη συζήτηση, αλλά να πω ότι εφόσον μιλάμε για κάτι που έχει να κάνει με την κουλτούρα, τα τρόφιμα και την επισήμανση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κάθε Ευρωβουλευτής έχει θέσεις για το θέμα αυτό. Και το θέμα αυτό ε, ε, είναι κάτι το οποίο θα έχει σημασία για 490, ε, για 490 εκατομμύρια πολιτών. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Ακόμα είμαι αισιόδοξη, ακόμα συνεχίζω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμούς. Ε, όλοι ε, θα πρέπει να κινηθούμε ο ένας προς τον άλλο, να επιδείξουμε ευελιξία για να βρούμε συμβιβασμού, του οποίου να μπορούν να υποστηρίξουν όσο γίνεται περισσότερε πολιτικέ ομάδε. Κύριε Πρόεδρε, ένα πράγμα θέλω όμω να πω με βάση τη συζήτηση που είχαμε σήμερα και με βάση τις πολλές συζητήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια στο Κοινοβούλιο. θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια εντελεχής έρευνα σχετικά με το τι κάνει τους πολίτες να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Τι μέσα μπορούμε εμείς οι πολιτικοί να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε συγκεκριμένη συμπεριφορά από τους καταναλωτές. Τι είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών, διότι όλοι μας θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους πολίτες ώστε να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για τους, για τους ίδιους. Αλλά τι χρειάζεται. Μερικοί θεωρούν ότι αρκούν οι πληροφορίες και ότι ο, ο καταναλωτής ε, ερμηνεύει τις πληροφορίες αυτές. Άλλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται καθοδήγηση ο καταναλωτής, ότι πρέπει να, φάει, πρέπει να του πούμε ότι πρέπει να φάει περισσότερα από αυτά και λιγότερα από αυτά τα προϊόντα. εμείς ε, σκεφτόμαστε τι είναι καλύτερο για τους εαυτούς μας και πώς φερόμαστε εμείς, ε, πώς ψωνίζουμε εμείς τα προϊόντα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνουν έρευνες σχετικά με το τι απαιτείται ώστε να φέρονται με συγκεκριμένο τρόπο οι καταναλωτές. Εμείς ως, ως πολιτικοί θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο τι μέσα λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας. Εν αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχω συγκαλέσει συνάντηση στις 2 Φεβρουαρίου και στις 10 Φεβρουαρίου για τους σκιώδεις εισηγητές. Και προτείνω να κάτσουμε πολύ συγκεκριμένα να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς για τα θέματα που συζητήσαμε. Μερικοί συμβιβασμοί θα είναι εύκολοι, μερικοί συμβιβασμοί νομίζω θα απαιτήσουν περισσότερη προσπάθεια, αλλά το εξή άκουσα σήμερα, ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι διατεθειμένοι να ε, εργαστούν με συμβιβαστικό πνεύμα και εμεί που δεν ε, αντιπροσωπεύουμε την πλειοψηφία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πολιτική πραγματικότητα. Η 23 Φεβρουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα και ρώτησα την Κατρίν σχετικά με τι άλλε επιτροπέ ε, και οι άλλε επιτροπέ, στο σημείο με εμά, δηλαδή συζητάνε τι τροπολογίε. Ε, η ε, Επιτροπή ΕΝΒΗ δεν έχει προχωρήσει, έτσι λοιπόν μπορούμε να επηρεάσουμε ακόμα τις εξελίξεις. Δεν έχω συζητήσει ακόμα με την ΕΝΒΗ τι θεωρεί η δική μα Επιτροπή, διότι δεν ήξερα τι ακριβώ θα έπρεπε να τη πω. Σας ευχαριστώ πάντως για τις πολλές παρατηρήσεις και προσβλέπω στη συνέχεια της συζήτησης τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κρίστελ Σάλτεμος, ε, που ηγήθηκε με τόσο στένο της διαδικασίας αυτή και που είναι τόσο ανοιχτή προσυζήτηση. Ε, συνάδελφοι, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και επιτρέψτε μου ε, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο θέμα αυτό, δεδομένη της απουσίας τη κυρία Χέτ. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, ακούσαμε πολλέ συνεισφορέ και έχουμε υποβάλει σχεδόν τι τριπλάσιε τροπολογίε από την επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή στο τέλος του πακέτου σας βλέπετε και μία ε, γραφική τροπολογία του κυρίου ε, Κρότσμαν. Μήπως λοιπόν θα σχεδιάσετε εσείς ε, νέα προγράμματα κύριε Κρότσμαν. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και ε, αυτή τη στιγμή εκεί βρισκόμαστε. 23 Φεβρουαρίου μάλλον θα ψηφίσουμε. Αυτό βέβαια ε, εξαρτάται και από τις εργασίες τη Επιτροπή ΕΝΒΗ, αλλά αυτό, αυτό είναι το σχέδιο. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο ε, θέμα μας. Βλέπω ότι αρκετοί αποχωρούν. Σας παρακαλώ. Όσοι δεν μείνετε για την επόμενη σημαντική συζήτηση να εγκατελείψετε την αίθουσα ήσυχα διότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην τέταρτη ανταλλαγή απόψεων για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, η συγητή μα είναι ο κύριο Σφαπ και νομίζω ότι είναι εδώ, ότι είναι παρόντε και οι περισσότεροι σκιώδει εισηγητέ. Ε, Αντρέα, να δώσουμε ένα λεπτό στον κόσμο να αποχωρήσει για να ε, έχουμε ησυχία πριν πάρει το λόγο και να αλλάξουν βάρδια οι παρευρισκόμενοι. Uh, uh Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Όσοι δεν θέλετε να παραμείνετε στην αίθουσα για την επόμενη συζήτηση, αποχωρήστε ησύχως. Περνάμε στην τέταρτη ανταλλαγή απόψεων λοιπόν για τα δικαιώματα καταναλωτών. Αυτή η οδηγία που είναι ένα από τα πιο σημαντικά που έχουμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί του παρόντος. Ο κύριος Σβάμπ θα αγηθεί τη συζήτηση. Ο κύριος Ντέφα δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Η κυρία Σάλτε Μόσε θα τον καλύψει, έτσι δεν είναι. Ο κύριος Ρόσχορ είναι εδώ. Η κυρία Τούρνεν είναι εδώ. Ήλαν Τριανταφυλλίδης. Α, δεν είναι εδώ. Ήταν όμως εδώ μέχρι πριν από λίγο. Θα δώσω το λόγο στους εισηγητές και σε όποιον άλλον θέλει να μιλήσει και η Επιτροπή εκπροσωπείται. Ο κύριος Κωνσταπέτρης είναι εδώ. Θα σας δώσω το λόγο στο τέλος για να σχολιάσετε κι εσείς. Ωραία. Και ο κύριος Κρέσπο βέβαια είναι πάντα εδώ. Λοιπόν, κύριε Σβάμπ, τέταρτη ανταλλαγή απόψεων. Ποια κατεύθυνση ακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τον ίδιο αστερισμό ε, σκιωδών εισηγητών με την προηγούμενη συζήτηση που επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια είναι διαφορετικό το θέμα μας εδώ. Πολύ σωστά αναφέρατε κύριε Πρόεδρε ότι πρόκειται για την τέταρτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι η συζήτηση που είχαμε μόλις πριν έδειξε ότι όταν είναι περισσότερες οι γνώσεις είναι και πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Ελπίζω λοιπόν ε, ο χωρισμός της συζήτησης σε κεφάλαια να ανεβάσει το επίπεδο της συζήτησης. Καταρχήν, για τους συνεδέρφους που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καλά το θέμα αυτό, να κάνω μια σύντομη παρουσίαση η κυρία Ρέντινγκ θα είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό στο μέλλον και στην ε, ακρόασή της ε, κατέστησε σαφές ότι είναι υπέρ της εναρμόνισης ε, της εσωτερικής αγοράς διότι πιστεύει ότι για παράδειγμα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών εάν δεν είναι στόχος της εσωτερικής αγοράς η εναρμόνιση τότε αυτό αποτελεί αυταπάτη. Ε, στοχεύει στην ε, στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ε, εισηγητή και τους σκιώτους εισηγητές της Επιτροπής μας. Είμαι αισιόδοξο ότι τα δύσκολα θέματα που έχουμε μπροστά μα θα μπορέσουμε ε, να τα ε, προχωρήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα η ακρόαση του κ. Ντάλι έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα μεγάλα και μικρά κράτη-μέλη. Τα μεγάλα κράτη-μέλη δεν κινδυνεύουν από τον ε, κατακαιρματισμό των ε, νομοθεσιών, ενώ τα μικρά κράτη-μέλη έχουν σαφώς τη θέση ότι αν δεν πετύχουμε ένα ελάχιστο καταναλωτικό νομοθεσία νομοθεσίας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι θα μειωθεί το επίπεδο στα μικρά κράτη-μέλη και δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να τα τροφοδοτήσουν τις μικρές αγορές. Να σας παρουσιάσω τις δικές μου σκέψεις για την ε, περαιτέρω ε, επεξεργασία του θέματος. Ε, το κεφάλαιο 5, με το οποίο θα, στο οποίο θα συγκεντρωθούμε σήμερα, επικεντρώνεται στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Απαγορευμένες ρήτρες στο καταναλωτικό δίκαιο της Ευρώπης. Η Κομισιόν προτείνει δύο διαφορετικούς καταλόγους, μία μαύρη λίστα με απαγορευμένες ρήτρες, ρήτρες που απαγορεύονται σε όλη την Ευρώπη και μία γκρίζα λίστα με ρήτρες οι οποίες πιθανώς να είναι εις βάρος του καταναλωτή. Πρόκειται για ένα σύστημα πλήρους εναρμόνισης. Με την βοήθεια της Επιτροπολογίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει σε όλη την Ευρώπη τη δυνατότητα να εισαχθούν ε, αλλαγές σε όλη την Ευρώπη. Στόχος των κρατών μελών κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο αλλά και εδώ στο Κοινοβούλιο Τα κράτη-μέλη θέλουν ευελιξία στην ομοθεσία τους. Ε, ζητούν λοιπόν ε, η αρχή αυτή να εφαρμόζεται και στο κεφάλαιο 5. Γι' αυτό υπάρχει επιφύλαξη απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν που εισάγει γενικές ρήτρε. Από την άλλη όμως, πιστεύω ότι μπορούμε να σκεφτούμε το θέμα μήπως Υπάρχουν ενιαίες αρχές που θα πρέπει να εισαχθούν στο καταναλωτικό δίκαιο σε όλη την Ευρώπη. Μήπως υπάρχουν πρακτικές οι οποίες θα πρέπει γενικά να τιμωρούνται. Πιστεύουμε λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τον μαύρο κατάλογο που ε, προτείνει η Επιτροπή. Είμαι ευγνώμων για τις ε, προτάσεις που άκουσα από διάφορες ε, ενώσεις καταναλωτών και άλλες που είναι διατεθειμένες να εξετάσουν τη στρατηγική αυτή και που ενδεχομένως να μην έχουν ακόμα σαφείς θέσεις. Πιστεύω ότι συμφωνούμε ότι και στο θέμα δεν θέλουμε επιτροπολογία στο ευαίσθητο αυτό θέμα για τους καταναλωτές. Μετά από 60 χρόνια Ευρώπης πιστεύω ότι υπάρχει κάποια συνοχή πια στην Ευρώπη που θα μας επιτρέψει μέσω πρόθεσμα, ίσως όχι τα επομενα 2 2-3 χρόνια, να απαγορεύσουμε συγκεκριμένες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη. Παράδειγμα, στις ε, για παράδειγμα να σας δώσω ε, την ε, να σας δώσω το παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται ο πολιτής λόγω σοβαρής αμέλειας να εξαιρείται από την ευθύνη, από την ευθύνη του να απαλλάσσεται από την ευθύνη του. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει τέτοιοι κανόνες να εισαχθούν ε, στη νομοθεσία των κρατών μελών ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν ε, να οδηγήσουν τους παραγωγούς σε αλλαγή των εμπορικών τους πρακτικών. Θέλουμε να ενισχύσουμε το δίκαιο των καταναλωτών και θέλουμε να αποφύγουμε, να απαγορεύσουμε τις ερήτρες που είναι εις βάρος των καταναλωτών. Των καταναλωτών. Κύριε Πρόεδρε, αυτές είναι οι βασικές μου σκέψεις για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι για το κεφάλαιο 5 μπορούμε να πούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η εναρμόνιση είναι ή όχι. Το θέμα είναι σε ποιους τομείς η πλήρης εναρμόνιση ωφελεί όχι μόνο την εσωτερική αγορά αλλά και τους καταναλωτές. Ελπίζω ε, να καταλήξουμε σε μια πρακτική λύση. Προσβλέπω στη συνέχεια τη συζήτηση ε, και να σας πω για το χρονοδιάγραμμα ότι μετά από την συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας θα ε, συνοψίσω τις θέσεις των συναδέρφων σε ένα έγγραφο το οποίο θα στηρίζεται στο έγγραφο της συναδέρφου Αρλίν Μακκάρθη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Η Σκιώδης, η κυρία Σαλεμόζα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα εκ μέρους της ε, Εύελιν να απολογηθώ για την απουσία της σήμερα. Δεν θα μιλήσω τόση ώρα όσο μίλησα για το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα τρόφιμα, διότι απλά δικαθιστώ την Εύελιν. Έχουμε ανησυχίες, ε, αυτό δεν θα σας εκπλήσει, σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση και στο κεφάλαιο 5. Ανδρέας, ανέφερε κάποια από τα προβλήματα που θα μπορούσαν να εμφανιστούν. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος να ακολουθήσουμε. Ε, ο Νορβηγός διαμεσολαβητής για τους καταναλωτές ε, μας ε, προειδοποιεί κατά κάτι τέτοιου. Τούτου λεχθέντος όμως ε, θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένας μαύρος κατάλογος, να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θέλουμε τις συγκεκριμένες ρήτρες, συμβατικές ρήτρες. Να πούμε δηλαδή ότι αυτές οι πρακτικές είναι σε όλη την Ευρώπη αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το θέμα είναι θα προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα, δηλαδή θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να μπορεί να προχωρήσει πιο πέρα ώστε με βάση την κουλτούρα, τις παραδόσεις, ε, τις νομοθεσίες των ε, κρατών μελών Εμείς θέλουμε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα, να θεσπίσουν δικού του κανόνες. Δεν πιστεύουμε ότι η πλήρης εναρμόνιση είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, η μαύρη λίστα είναι ενδιαφέρον τρόπος, ε, αρκεί να μην είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή. Αυτά είχα να πω σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάλτε Μόσε, ο κύριο Ροσφόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή που μας υπενθύμησε τα όσα ήδη έγιναν υπό την αιγίδα σας στις πρώτερες συνεδριάσεις. Πάντα αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ναι, η αποδοχή της αρχής της μέγιστης εναρμονίσεως υπό τον όρο ότι αυτό θα είναι κάτι που δίνει προστιθέμενη αξία, αλλά όχι να οδηγεί σε κάτι αρνητικό για να πάμε κατευθείαν στο σκοπό του κεφαλαίου, η μέγιστη εναρμόνιση. Εάν θέλουμε να συμφωνήσουμε επί των συγκεκριμένων ορισμών της ρήτρα της καταχρηστικής δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Αν θέλουμε να συμφωνήσουμε επί του, των συνεπειών αυτής της ρήτρα, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αν πούμε ότι σε περίπτωση αμφιβολιών τα ωφέλη θα πρέπει να είναι υπέρ του καταναλωτού και εκεί συμφωνούμε τούτων των σημείων λεκθέντων καταλήγουμε στην ε, πρακτική προσέγγιση. Οι δύο συνάδελφοί μου αναφέρθηκαν στο θέμα των καταλόγων. Όσον αφορά αυτό το θέμα, μαύρος κατάλογος, μαύρη λίστα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να έχουμε ένα κατάλογο ο οποίος να μπορεί να ισχύει σε όλες χώρες της Ένωσης. Τίθεται όμως το εξή. Αυτή η λίστα και αυτή και η γκρίζα λίζα εντάσσονται στο πλαίσιο της μέγιστης εναρμόνισης ή αντίθετα συνεπάγεται ότι αυτό που δεν είναι στη μαύρη λίστα δεν θα προσθεθεί, δεν θα, δεν θα το εφαρμόσετε κάτι μέλη. Σε αρκετά κάτι μέλη ε, το υπενθύμησε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο Ευρωπαϊκό, κράτο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσον αφορά τη μέγιστη εναρμόνιση δεν μπορεί να προσθέσει κάτι ένα κράτος. Υπάρχουν χώρες σήμερα που δεν έχουν μαύρη λίστα και στις χώρες εκεί ε, υπάρχει σημαντική πρόοδος. Και υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ πλήρεις καταλόγους ανάλογα με τα διάφορα θέματα. Αν πάρω τη χώρα μου, τη Γαλλία, στον τομέα των ε, κινήτων υπάρχουν 20 ρήτρε παράνους αφορούν ε, τις σχέσεις με τους ενοικιαστές. Και θεωρούμε ότι αυτή η εξάρτηση που υπάρχει μεταξύ ιδιοκτήτου και αυτού όσον αφορά τη στέγαση στην παρούσα κρίση είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαφέ ότι στον παρόντα ορισμό των καταλόγων όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί δεν βρίσκουμε αυτού του είδου τι πληροφορίε και τι λεπτομέρειε. Τέλο, αυτό που θα θέλαμε όλοι θα ήταν να υπάρχει αυτή η μαύρη λίστα και η δυνατότητα σε κάποιες χώρες να υπάρχουν και συμπληρωματικοί κατάλογοι που είναι κάτι κεκτημένο για τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν μιλάμε τώρα στη μέγιστη εναρμόνιση αφορά τον ορισμό των καταλόγων αυτών. Το άρθρο 32, προσέξτε, στο άρθρο 32 ε, διευκρινίζεται υπό ποιου όρους ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να επικαλεστούν μια ρήτρα καταχρηστική χωρίς αυτή να συμπεριλαμβάνεται στην μαύρη, στη θεά λίστα. Και αυτή είναι η αναφορά στις γενικές αρχές όπως αποκαλείται όπως είναι η διάταξη εισάρρωσης. Ε, εγώ ανησυχώ. Το άρθρο αυτό 32 είναι σαν να θέλει να ανακτήσει, να καλύψει όσα δεν καλύπτονται τις δύο καταλόγους. και ίσως να δημιουργεί κάτι που είναι και δεν είναι ασφάλεια δικαίου. Διότι ο δικαστής, οι εθνικοί δικαστές των κρατών μελών θα πρέπει να ερμηνεύσουν τις γενικές αρχές πέρα από τις δύο λίστες. Αν γίνει αυτό, μήπως καταλήξουμε κάπου που αντί να βοηθήσει και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εναρμονισμένους ορισμούς οδηγήσει σε κάτι πολύ ευμετάβλητο που θα εξαρτάται από την ερμηνεία των δικαστών κάθε κράτους. Έχουμε πολλά ερωτηματικά επ' αυτού. Συμφωνώ με τον κ. Σβάμπ. Η επιτρολογία φαίνεται κάτι παράξενο για κάτι τέτοιο για την προσέγγιση στην ανθρώπινη πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή του καταναλωτού. Αυτό αντιπροσωπεύουν αυτές οι λίστες. τίθενται και άλλα ερωτηματικά. Υπάρχουν σημεία που αφορούν άλλα άρθρα. Δεν ξέρω αν παρευθείς θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη. τη ρήτρα που είναι αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης σε σύγκριση με τις προκαθορισμένες τυπικές διατάξεις που υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη. Επέκταση της εφαρμογής αυτών των ρητρών, των καταχρηστικών, στις, που επεκτείνονται και καλύπτουν και τις ρήτρες που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης εξειδικευμένης. Αυτό είναι λεπτομέρεια, πρέπει να συζητηθεί. Ως έχει το κείμενο του σχεδίου οδηγίας, η μη συμπερίληψη άμεση αυτών των ρητρών που είναι αντικείμενο εξειδικευμένη διαπραγμάτευσης στις γενικές αρχές, ίσως οδηγήσει σε λύσεις που θα κατακριθούν από διάφορες επιχειρήσεις. Χρειάζεται συντονισμός και με την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που θα μπορεί να πει κάποια πράγματα πάνω σε αυτά. Και το άρθρο 30 αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογή αυτών των ρητρών. Έχουμε πολλά και στο άρθρο 31 που είναι αρκετά ενδιαφέρον αναφέρεται στις ε, υποχρεώσεις διαφανείας σε αυτές τις συμβατικές ρήτρες. Χρειάζεται εύληπτη γλώσσα να χρησιμοποιείται και διαφανής και λέει ότι τα κράτη-μέλη απέχουν από το να επιβάλλουν η απέτηση στο εδάφιο 4 το άρθρου 31 δεν επιβάλλουν επίσημες απαιτήσεις, τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διατύπωση των συμβατικών αυτών ρητρών ή πώς αυτές τίθεται στη διάθεση του καταναλωτού. Και εδώ δημιουργούνται ερωτηματικά έναντι κάποιων καταναλωτών. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να δεχτούμε την αρχή της μέγιστης εναρμονίσεως πάνω σε πλαισιωμένα ζητήματα. Χρειάζεται να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, κυρίως όσον αφορά τις λεπτομέρειες όσον όλων αυτών των ρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλές οι παρατηρήσεις όλες που κάνατε. Και βέβαια πρέπει να δούμε και την οδηγία της εμπορικές πρακτικές. Η κυρία Τιούρινεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να έρθω λιγάκι στο τελευταίο σημείο του κύριου Ράσφαλ και τρία πράγματα έχω να πω για αυτό το κεφάλαιο σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ποιε συμφωνίε καλύπτονται και ποιε δεν καλύπτονται. Για μένα δεν είναι ξεκάθαρο. Και αυτό έχει να κάνει και με τι ατομικέ ε, διαφορέ. Δεύτερον, είναι εύκολα κατανοητό. Και τρίτον, εναρμόνιση και τι προσέγγιση ακολουθούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτα απ' όλα, για το ποιε συμφωνίε καλύπτονται και ποιες όχι, ποιες συμβάσει δηλαδή. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα μένουν απ' έξω ετομικές συμφωνίες γιατί όπως είπε και ο κ. Σούρφαλ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής δεν μπορεί να επηρεάσει τη συμφωνία και τον τρόπο με τον οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Εκεί μπορεί να οδηγηθούν σε ένα ατομικό ε, συμβόλαιο, συμφωνία και να μην καλύπτονται. Πρέπει λοιπόν εδώ να βρεθεί μια διέξοδο. Επίση, και αναφέρθηκε και αυτό, υπάρχουν και συμβάσει για την ενοικίαση διαμερισμάτων. Καλύπτεται αυτή η περίπτωση ή όχι. Η Επιτροπή επιτροπη ισω θα μπορούσε να μα το πει αυτό. Για μένα δεν είναι ξεκάθαρο. Με έχουν ρωτήσει διάφοροι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεν ξέρω τι να απαντήσω ακριβώ. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου απαντήσει. Το άλλο γι' αυτό είναι ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς εύκολα να διαβάσει τους όρους της σύμβασης. Εδώ λέει στο άρθρο 31 ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι αναγνώσιμο και τι όχι. Είναι αυτή εδώ η οδηγία που αποτελεί την απόρρια της αναρμονημένης προσέγγισης να καθορίσει το τι είναι αναγνώσιμο και τι όχι. Και είναι αδύναμη αυτή η οδηγία εδώ, γιατί λέει ότι εξαρτάται από τις επιχειρήσεις και από τους πολιτές οι οποίοι θα αποφασίσουν τι διατύπωση θα ακολουθήσουν. Το μέγεθος, διατύπωση, όλα. Οπότε και εδώ υπάρχει ένα κάποιο πρόβλημα για το ποιος τελικά καθορίζει το τι είναι ξεκάθαρο, τι είναι κατανοητό, τι είναι ευανάγνωστο. Και αν δεν είναι ευανάγνωστο, τότε τι θα γίνει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να λύσουμε, να απαντήσουμε. Αν με ρωτήσετε εμένα, εννοείται ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι υπέρ του καταναλωτή. Ότι δεν δεσμεύεται πια από τη συμφωνία. Και το τελευταίο μου είναι ότι η πλήρης εναρμόνιση με μαύρη λίστα, γκρίζα λίστα είναι κάτι που δεν βοηθάει. Γιατί το ερώτημα είναι, δεν υπάρχουν τόσο διαφορετικές συνήθειες και διαφορετικές προδιαγραφές στα κράτη-μέλη που να πρέπει να επιτρέπουμε επιπλέον από τον κατάλογο αυτό, τον κοινό που θέλουμε να έχουμε. Έτσι νομίζω. Θα προτιμούσα λοιπόν μια προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης στο κεφάλαιο αυτό. Αν τώρα η επιχείρηση θέλει να πουλάει σε ολόκληρη την Ευρώπη, αρκεί να πετύχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο δικαιωμάτων και να τα θεωρήσει σαν ε, γενικό κανόνα για αυτή την επιχείρηση. Εδώ εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Αν έχουμε δηλαδή τις ελάχιστες προδιαγραφές. Μπορεί κάποιος να βάλει ψηλές προδιαγραφές, δεν υποκλείεται. Και για να συνοψίσω. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και πραγματικά αυτό το θέμα της εναρμόνισης. Κύριε Σβάμπ, για συνοψίστε μας τις δικές σας απόψεις, γιατί το συζητήσαμε λίγο, αλλά δεν έχω πάρει μια σαφή απάντηση όσον αφορά το επίπεδο αναρμόνισης που επιθυμείτε εσείς. Ευχαριστούμε για τα ξεκάθαρα σημεία που θέσατε. Ο κύριος Βίλερ τώρα. Βίλεν. Ευχαριστώ. Είμαστε σε μια τέταρτη ανταλλαγή απόψεων για την οδηγία αυτή και είναι καλό που αποφασίσαμε να εμβαθύνουμε κάπως στη συζήτηση ανακεφάλαιο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να περάσουμε από το επίπεδο της συζήτησης στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Γιατί πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για κάποια στοιχεία κλειδί. Το ανέφερε και ο κύριος Φαμπ. Για παράδειγμα το θέμα της πλήρους εναρμόνισης. Είναι ένα επίμαχο θέμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε. Όσον αφορά το κεφάλαιο 5 που αναφέρεται στους όρους της συμφωνίας, εδώ είμαι κάπως πιο επιφυλακτικός για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω μελετήσει την πρόταση της υπηρεσίας της πολωνικής προστασίας των καταναλωτών. Έχουν εξετάσει εκατοντάδες συμβόλαια από πέρυσι και η υπηρεσία αυτή θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά πολλέ τέτοιε συμφωνίε, οι οποίε δεν είναι σωστέ, δεν είναι θεμητέ. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε και στη χώρα μου να αποκτήσουμε καλύτερε προδιαγραφέ συμφωνιών. Θέλω να ξέρω ποια είναι τα επιχειρήματα των ε, βουλευτών από τη Σοσιαλιστική Ομάδα, που ανέφερε συνάδελφο από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Όσον αφορά τώρα τις λίστες, την μαύρη και την κρύ, αν αποφασίσουμε για την αναρμόνιση του κεφαλαίου 5, τότε δεν χρειαζόμαστε πια τις λίστες αυτές. Δεν έχει πια νόημα. Είναι δύσκολο να έχουμε το κεφάλαιο χωρίς τις λίστες. χάνεται το νόημά τη η οδηγία. Πάντως συμφωνώ με τον συνάδελφο από την άλλη ότι δεν πρέπει να είναι κλειστή κατάλογη αυτή. Όχι, πρέπει πάντα να υπάρχει δυνατότητα να συμπληρωθούν οι λίστες αυτές με κάτι που θα προκύψει και η γκρίζα και η μαύρη λίστα. Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω τον κύριο Σβάμπ όσον αφορά τη διαδικασία επιτροπολογίας. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει νόημα η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής εδώ. Ευχαριστώ. Και Τελευταίος από τους κοιόδους, ο κύριος Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς πιστεύουμε ότι το κεφάλαιο αυτό της οδηγίας που συζητάμε σήμερα είναι ένα από τα πιο αδύνατα σημεία της όλης οδηγίας. Και αυτό γιατί η δημιουργία της μαύρης και της γκρίζας λίστας ανοίγει, όπως τα λέγαμε, τους ασκούς του αιώλου για το κοινοτικό δίκαιο. Και αυτό πολύ απλά γιατί το άρθρο 38, παράγραφος 2, δίνει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να κάνει χρήση του εθνικού δικαίου για να κρίνει κατά πόσο συμβατικές ρήτρε που συντάχθηκαν για γενική χρήση είναι καταχρηστικές ή όχι. Άρα παρόλο που θα υπάρχει η αρχή του κοινοτικού δικαίου, αυτή θα προσβάλλεται συνεχώς με υποθέσεις στα εθνικά δικαστήρια. Πώς προστατεύεται έτσι ο καταναλωτής. Η Επιτροπή έχει μελετήσει τι σημαίνει με, σε νομοθετικό όγκο η πιο πάνω δυνατότητα έχει υπολογίσει το νομοθετικό αλαλούν που θα δημιουργεί για το ποια ρήτρα θα ισχύει και σε ποια χώρα. Είναι με αυτόν τον τρόπο που θα επιτευχθεί η καθολική προστασία των καταναλωτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς πιστεύουμε ότι η πλήρης εναρμόνιση δεν πετυχαίνει την προστασία των καταναλωτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Στη δική μας αντίληψη αυτό δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο Πέραν το ότι απλά με αυτές τις δύο λίστες η οδηγία εναρμονίζει ένα με επίπεδο προστασίας για τις καταχρηστικές ρήτρες, τις καταχρηστικές συμβάσεις, επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους νομικά ισχυρούς οργανισμούς να αφισβητούν με νομικά μέσα τις καταχρηστικές ρήτρες και άρα να έχουν το πάνω χέρι στη σχέση τους με τους καταναλωτές. Με απλά λόγια, οι μεγάλες επιχειρήσεις που ελέγχουν την αγορά θα μπορούν ανα πάσα στιγμή σε κάθε κράτο μέλο, να αμφισβητούν την εφαρμογή αυτών των καταλόγων και άρα να διαμορφώνουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτές επιθυμούν. Πώς επιτυχάνουμε προστασία για τους μεμονωμένους καταναλωτές, πώς διασφαλίζουμε την επιβολή αυτών των ρητρών. Και επιπρόσθετα, το ζήτημα της πολιτικής πολυπλοκότητας του κειμένου με την υπερβολική χρήση παραπομπών δημιουργεί επικοδομητικές ασάφειες. Αυτές οι ασάφειες δεν πρόκειται να τύχουν εκμετάλλευση από τους καταναλωτές, αλλά μάλλον οι επιχειρήσεις θα τις αξιοποιήσουν στο ΕΠΑΚ. Μια πολύ βασική αρχή πρέπει να τηρηθεί σε οποιαδήποτε νομοθεσία καταπιάνεται με το ζήτημα προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη πρέπει να είναι άθικτη. Ωστόσο, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποτελεί όπλο για τη συνεχή μείωση του επίπεδου προστασίας των καταναλωτών. Αυτή είναι η θέση μας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Uh, um, λοιπόν, για άλλους που θέλουν να πάρουν το λόγο, και κ. Χαουνό, κυρία Ράπτη και ο κ. Κουπάκης. Θέλει και άλλος να πάρει το λόγο. Ο κ. Χουάν Νοκ, καταρχάς. Πρόεδρε, όπως και πολλοί συνάδελφοι είπαν σε αυτή την Επιτροπή και εγώ έχω επιφυλάξει όσον αφορά την επιλογή της Επιτροπής όσον αφορά τη μέγιστη εναρμόνιση έτσι θα πάγωνε κάθε προπτική προόδος όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, αλλά επίση θα μειωθούν κάποιε εθνικά επίπεδα προστασία. Όσον αφορά το πέμπτο κεφάλαιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τη μέγιστη εναρμόνιση είναι ότι θα οδηγούσε να στερηθούμε κάθε δυνατότητα ταχεία αντιδράσεω. Ακόμα και αν οι τρόποι κατανάλωση εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα, και άρα υπάρχει κίνδυνος να ξανεμφανιστεί μια νέα ρήτρα καταχρηστική. Η πρώτη οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα προσαρμογή της ε, νομοθεσίας μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας, όμως το να ανανεωθεί η διαδικασία της επιτροπολογίας στο Κοινοβούλιο με θετικότερο τρόπο δεν κάνει τα πράγματα πιο διαφανή και πιο δημοκρατικά. Στην περίπτωση της Γαλλίας που γνωρίζω καλύτερα, ο κατάλογος των ρήτρων που, που θεωρούν καταχρηστικές ξεπερνά ήδη αυτά που εμφανίζονται στο παράρτημα 1. Ε, γι' αυτό ε, εγώ στα πλαίσια της οδηγίας είμαι υπέρ προσεγγίσεως μικτής. Ανάμεσα στα στοιχεία που ίσως ε, αποτελέσουν αντικείμενο μέγιστης εναρμονήσεως, υπό τον όρο ότι οι βελτιώσεις τα λάβουν χώρα, θα έθετα, τον ορισμό ή τους κανόνες που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, της δυνατότητας ανάκλησης. Ε, όμως δεν θα ήταν ευκταίο ότι δυνατόν να ερμονιστούν πλήρως οι διατάξεις όσον αφορά τις υποχρεώσει ενημερώσεως ή τις υποχρεώσεις που αφορούν τις καταχρητικές διατάξεις της ρήτρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν πιο πέρα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Uh, Mr. Ο κ. Πουπάκης. Το μικρόφωνο σας. Αναφορικά με το κεφάλαιο 5 της οδηγίας, στέκομαι κυρίως στο ζήτημα των καταχρηστικών ιτρών που ορίζονται σε αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή χωρίζονται οι συμβατικές ως καταχρηστικές σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη τη μαύρη που περιλαμβάνει πέντε μόνο περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται αυτομάτως σε κάθε περίπτωση καταχρηστικές, ενώ στη δεύτερη την κρή οι 12 περιπτώσεις, οι περισσότερες δηλαδή, τεκμέρονται σαν καταχρηστικές εκτός και αν ο έμπορος αποδείξει το αντίθετο. Δηλαδή περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει προστασία χαμηλότερου επίπεδου από αυτή την πρώτη κατηγορία. Ενδεικτικά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω τον κίνδυνο που ανέφερε ο κ. Βάπ στην αρχή, ότι σε αρκετέ χώρε, όπω και η ελληνική νομοθεσία η δική μα, περιλαμβάνει ένα μόνο κατάλογο χαρακτηριστικών ρητρών, οι οποίε είναι στο σύνολό του και υπό οποιασδήποτε συνθήκε καταχρηστικέ, σε αντίθεση με την πρόταση τη οδηγία. Και δεύτερον, ένα μόνο κατάλογο χαρακτηριστικών ρητρών, οι οποίε είναι στο σύνολό τη και υπό οποιασδήποτε συνθήκε όπω αναφέρουμε καταχρηστικέ. Επειδή λοιπόν η αρχή τη πλήρου εναρμόνιση θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί σε μερικά κράτη-μέλη η προστασία των κανοντών, καθώ δεν θα μπορούν να θεσμοθετήσουν επιπρόσθετα δικού του καταλογού και δεν θα μπορούν να προσθέσουν επιπλέον καταρχιστικέ ρήτρε στου καταλογού. Γι' αυτό ίσω θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνει μια εκτενής επεξεργασία των μαύρων και γκρίζων καταλόγων των κρατών μελών ώστε να γίνει ένας ενιαίος κατάλογος καταχρηστικών, δεύτερον να συμπεριληφθούν πρόσθετες από τις ήδη εγγυημένε που υπάρχουν, εγγυήσει που υπάρχουν στα περισσότερα κράτη. Διαφορετικά, σε αντίθετη περίπτωση, ίσως θα πρέπει να υπάρξει είτε ευελιξία στην εναρμόνιση, είτε ελάχιστη εναρμόνιση στα κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σε αρκετά κράτη-μέλη να πάμε πίσω από την προστασία που ήδη έχουμε θεσμοθετήσει σε αυτά τα κράτη. Ευχαριστώ. Κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πριν από όλα θέλω να πω ότι εύχομαι καλή επιτυχία και στη συνέχεια της δουλειάς και στον κύριο Σουάπ και στους α, σκιώδες εισηγητές γιατί είναι μια καθαρά δύσκολη δουλειά και νομίζω ότι χρειάζεται κουράγιο για να συνεχίσουν. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για μας στην Ελλάδα και ο κύριος Κουπάκης, ο προηγούμενος ομιλητής, είναι από την Ελλάδα, ε, από διαφορετικό κόμμα από αυτό στο οποίο ανοίγω εγώ και έχει σημασία ότι θα με ακούσετε να συμφωνώ. Να συμφωνώ λέγοντας ότι το ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης για μας στην Ελλάδα είναι σημαντικό και είναι σημαντικό γιατί έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όσον αφορά το θέμα της μαύρης και της γκρίζας λίστας, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από αυτές τις λίστες. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα πριν φτάσουμε στο επίπεδο της μαύρης και γκρίζας λίστας. Ε, και ένα τελευταίο έχει να κάνει με το πόσο εύληπτα είναι όλα αυτά για τον καταναλωτή. Διότι συνήθως, ακόμα και αν έχουμε την τέλεια νομοθεσία, αυτή μένει στα χαρτιά και είναι ελάχιστοι οι καταναλωτές που εποφελούνται από την νομοθεσία. Άρα ένα επιπλέον στοιχείο είναι η νομοθεσία στην οποία θα καταλήξουμε και που ελπίζω να είναι καλύτερη και προς όφελος κυρίως των καταναλωτών θα πρέπει να φτάνει ως δικαίωμα σε αυτούς και να τους κάνουμε πιο εύκολο να την χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό που είπατε για εφαρμογή ε, είναι κάτι που το, στην αξιολόγηση συνεπιών το κουβεντιάσαμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα το εξετάσει και επανέρχομαι στη δουλειά που κάναμε στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία, την υλοποίηση οδηγίας. Υπάρχει έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Τον κύριο Κωνσταπέτρη της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλό να μοιραστεί κάποιες σκέψεις μαζί μας και ο κύριος Κρέσπο αν θέλει να μας ενημερώσει για την πρόοδο στο Συμβούλιο και μετά θα καλέσω τον κύριο Σβάπ να συνοψίσει. Ο κύριος Κώστα Πέτρη έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Uh, Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα. Δείχνει την πρόκληση που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντιμετωπίζουν τώρα ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ε, συμφερόντων του να έχουμε πλήρως εναρμονισμένους κανόνες για τους αθέμητους όρους των συμβάσεων και να καταλήξουμε σε κοινούς κανόνες για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τις εταιρείε να μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο πλαίσιο σε διασυνοριακές συναλλαγές και εμπόριο. Υπάρχει κέρδος, κάτι μπορεί να κερδίσουμε από όλα αυτά. Και κάτι άλλο που υπόθηκε εδώ είναι να το συσχετίσουμε αυτό με ευελιξία στα κράτη-μέλη όταν αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με καταχρηστικές ρήτρε στις συμβάσεις. Τι επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επέλεξε να κάνει μια προσπάθεια να πετύχει την ισορροπία που έλεγα. Πώς. Πρώτον, καθορίζοντας κάποιους όρους που θα απαγορεύονται, κάποια πράγματα που θα απαγορεύονται εν πάση περιπτώσει. Και χαίρομαι που κάποιοι το υποστήριξαν σαν ιδέα. Και για λόγους ευελιξίας θέλαμε να έχουμε και κατάλογο με αθέμητους όρους Απ' την άλλη θέλαμε για να βρούμε μια ισορροπία να επιτρέψουμε στα εθνικά δικαστήρια να υπάρχει επαρκής ευελιξία όσον αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις εφαρμόνοντας τη γενική ρήτρα του άρθρου 32 της προτάσεως. Έτσι θα συμπληρωνόταν οι σαφέστατοι κανόνες των καταλόγων. Δεύτερον, για να απαντήσουμε στην επίκριση που ακούστηκε ότι η πλήρης εναρμόνιση είναι άκαμπτη όταν προκύπτουν νέες καταστάσεις. Γι' αυτό προτείναμε ρήτρα περί επιτροπολογίας. Να συμπεριληφθεί αυτή η ρήτρα. Ακούστηκαν πολλές επικρίσεις σήμερα σχετικά με αυτό αλλά πρόθεσή μας, έχετε υπόψη, ήταν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ευελιξία. Να είναι πιο εύκαμπτη η διαδικασία τροποποίησης των ληστών αυτών. Να σας υπενθυμίσω ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας χρειάζεται επικαιροποίηση της προτάσεως για να ληφθούν υπόψη αλλαγές των διαδικασιών. Η διάταξη περί πρέπει να αντικατασταθεί από την ανάθεση πράξεων, εκχώρηση πράξεων, τη σχετική διάταξη προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί σχετικά με αυτό και να δει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. Αυτό είναι το υποβαθρό. Πιστεύουμε ότι εξασφαλίζεται επαρκής ευελιξία κάποια σχόλια σχετικά με τα ερωτήματα που ετέθησαν από διάφορους βουλευτές σήμερα. Οι όροι που είναι αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης εξαιρούνται από την πρόταση. Η νομοθεσία των κρατών μελών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το τι είναι αθέμητο, τι λαμβάνεται υπόψη στα ατομικά, στα ατομικές συμβάσεις. Θέλαμε να είναι εστιασμένο ο κανονισμό. και γι' αυτό αφήσαμε αυτά απ' έξω και τα κράτη-μέλη ρυθμίζουν, ε, διατηρούν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τι ατομικέ συμβάσει και του σχετικού όρου στα πλαίσια εθνική νομοθεσία. Υπάρχει και ρήτρα διαφύλαξη. στο άρθρο 30 παράγραφο 2. Δεν μπορεί ο να ξεφύγει εύκολα. Αν επηρεάσει ο καταναλωτής έναν όρο, το, το 32 βλέπει ένα τυποποιημένο το υπόλοιπο τμήμα της συμβάσεως. Και εν τη αυτή περιπτώση καλύπτεται από την προστασία που προβλέπει η πρότασή μας. Τέλος, οι συμβάσεις μισθώσεως πραγματικά καλύπτονται από το συγκεκριμένο κεφάλαιο της πρότασης. Uh, um, Σας ευχαριστώ πολύ με ενδιέφερε το ότι θέλετε να δώσετε στα δικαστήρια 100 μελών ευελιξία να ερμηνεύσει συγκεκριμένε υποθέσει. Κατά πόσο αυτό ταιριάζει με τι εναρμονισμένε διατάξει, δεν ξέρω. ο κ. Βάμπη το θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Εγώ δεν είμαι δικηγόρο και δεν ξέρω, ίσω ακούσουμε κάποια εξήγηση εν ευθέτω χρόνο. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε τι πρόσφατε υποθέσει για θέμητε εμπορικέ πρακτικέ, τη σχετική οδηγία. Κάποια θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι είναι αντικείμενο του πρωτοδικίου που σταμάτησε τους Βέλγους από το να επεκτείνουν τις διατάξεις της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, διότι θεωρήθηκε ότι αυτό αφήνει εκτός εθνική νομοθεσία, εξαιρεί εθνική νομοθεσία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που συζητούμε τώρα. Υπάρχει κάποια αναλογία εκεί που σίγουρα ο εισηγητής μα θα θέλει να εξετάσει. Κύριε Κρέσπο, θέλετε να μα ενημερώσετε εντάχει για την πρόοδο στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι οι συζητήσεις που άκουσα εδώ δεν ε, απομακρύνονται και πολύ από τις ζητήσει που έχουμε στο Συμβούλιο. Θέλω πάντως να σας πω ότι μετά από την τελευταία συζήτηση που έγινε εδώ στην Επιτροπή για το κεφάλαιο 4 της πρότασης, είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση του Συμβουλίου μεταξύ των Υπουργών, όπου συζητήθηκαν διάφορα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν και με προηγούμενες συζητήσεις που κάνατε εσείς εδώ. Ένα από τα θέματα αυτά είναι οι όροι ενός συμβολέου εξαποστάσεως, τα κεφάλαια 1 και 3 όπου οι περισσότερες χώρες στήριξαν τη διεύρυνση των ορισμών αυτών, ώστε να καλύπτονται και διάφορες περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται και να μην υπάρχει εκεί αθέμητος ανταγωνισμός. Για παράδειγμα, εφόσον χρησιμοποιούνται εξ αποστάσεως μέσα ή γίνεται μια προσφορά και διαπραγμάτευση γίνεται εκτός ε, κράτους. Επίσης, υπήρξε μια συμφωνία, οι περισσότερες χώρες το στήριξαν, την εναρμόνιση για 14 ημέρες για τα εξαποστάσεως ε, συμβόλαια και κοινέ προδιαγραφές για τέτοιες περιπτώσεις. Η ε, Το ότι αποκλείονται ορισμένε περιπτώσεις συμβάσεων, όπως συζητήθηκε και εδώ, συζητήθηκαν ιδιαίτερα οικονομικού χαρακτήρα συμβάσεις ή οικοδόμηση κατοικιών που πρέπει να αποκλείονται από τα κεφάλαια 2, 3 και 4. Και γενικά η πρόθεση είναι να μην καλύπτονται ε, οι κατασκευές νέων κτηρίων, αλλά ναι οι ανα... ανακαινήσεις. Νομίζω ότι πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίε που έχει αναλυθεί τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τα δικαιώματα του καναλητή και καλό είναι να προχωρήσουμε και να φέρουμε σε αίσιο πέρας την υπόθεση αυτή. Uh, um, Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, χρησιμότατες οι συνεισφορές τους. Να δώσω τώρα στον εισηγητή το λόγο για να συνοψίσει και να μας πει ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή η ανταλλαγή απόψε μου του συναδέλφου επί του κεφαλαίου 5 ήταν πολύ επικοδομητικέ. Ευχαριστώ όλου για τι πολύ ε, θετικές θετικέ τους. του. Ε, ανέλησαν πράγματα. Όπως σα είπα, όλα αυτά τα σημεία θα τα συμπεριλάβω στο έγγραφο εργασία μου αυτά που ακούστηκαν και τις διάφορες κρίσεις και ευχαριστώ εκ των προτέρων τη γραμματεία που, για τη βοήθειά τη. Όπως αναφέρθηκε αυτή δεν είναι εύκολη δουλειά αλλά με ικανοποιεί πολύ αυτή η δουλειά να συνοψίσω σύντομα. Θα πρέπει να προσέξουμε στον τομέα αυτών του δικαίου των καταναλωτών να μην υπερβάλλουμε όσον αφορά την εναρμόνιση. Ε, η πρόταση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, αλλά πιστεύω ότι σε πολλά σημεία θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μέτρο ώστε να εποφεληθούν οι καταναλωτές και να εφαρμοστεί σωστά από τα κράτη-μέλη. Ε, αγαπητέ Κυριάκο, συνάδελφε Τριανταφυλλίδη, Φυσικά θέλω υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή με την οδηγία αυτή. Ε, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το επιχείρημα της ε, προστασίας του καταναλωτή σε πολλά κράτη-μέλη δεν θα έλεγα ότι γίνεται αντικείμενο κατάχρησης, αλλά χρησιμοποιείται για να εμποδιστούν τροποποιήσεις στο εθνικό δίκαιο που είναι απαραίτητες. Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να πληρώσουμε κάποιο τίμημα και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην νομοθεσία των κρατών μελών. Ωστόσο, συμφωνούμε και νομίζω το έδειξε αυτό η συζήτηση ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό βαθμό ευελιξίας ώστε να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα οι προσαρμογές ε, ε, στην εσωτερική τους τάξη. Ωστόσο, οι καταναλωτές που επωφελούνται από την εσωτερική αγορά και το ε, ανέφερε αυτό ο Μάρκομ Χάρμπορ, Μην ξεχνάμε ότι με τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 και ε, ε, Ρώμη 1 θέλουμε τροποποίηση του σχετικού πλαισίου και έχουν γίνει σχετικές αποφάσεις στο Αρπενχόφ. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κάποιες ε, δυσκολίες, αλλά γενικά για το κεφάλαιο 5 μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε επιτροπολογία, ε, η επασύπτωση ανάθεση τη εκπόνηση τη νομοθεσία. δεν θέλουμε γκρίζα λίστα, φεά λίστα. Θέλουμε όμως να εξετάσουμε προσεκτικά και συγκεκριμένα μήπως στην μαύρη λίστα υπάρχει βάση να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες ε, να προσανατολίζονται σε αυτά που ήδη υπάρχουν στην νομοθεσία των κρατών μελών. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα απλά να σας δώσω μια γενική επισκόπηση, δεν ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες ε, του εγγράφου, ε, γι' αυτό δεν επικεντρώθηκα και στον Νορβηγό διαμεσολαβητή για τους καταναλωτές Άλλωστε οι Νορβηγοί δεν είναι καν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ε, γι' αυτό δεν ασχολήθηκα πολύ με το θέμα εναρμόνιση ναι ή όχι. Είπαμε θέλουμε στοχευμένη εναρμόνιση στου τομείς όπου έχει προχωρήσει η εσωτερική αγορά, ενώ στο μίσο που δεν έχει προχωρήσει η εσωτερική αγορά δεν θέλουμε πλήρη εναρμόνιση. Σα ευχαριστώ για τι παρεμβάσει σα. Ε, προτείνω, όπω πρότεινε και ο συνάδελφο ε, με του ε, σκιώδει να εκπονήσουμε έγγραφο εργασία, το οποίο ελπίζουμε στι αρχέ του Απριλίου να το έχουμε έτοιμο και κατόπιν να συζητήσουμε. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να καλέσουμε την Επίτροπο Ρέντινγκ στην ε, Επιτροπή μας μόλις ε, εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορούμε να έχουμε συζήτηση σχετική μαζί της. Εν μέρη έχει γίνει αυτό σε διμέρες επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στη συνέχιση της καλής συνεργασίας. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνεις και την ηγεσία σου από το θέμα. Να επενθυμίσω σε όλους, μέλη και συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, ότι αύριο το απόγευμα θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση από αυτού του θέματος μέσω βιντεοδιάσκεψης. Θα είναι η πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω που θα κάνει κάτι τέτοιο το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν κάποιο εθνικό κοινοβούλιο το έχει κάνει αυτό. Συγχαίρουμε την Γαλλική Εθνοσυνέλευση που το κάνει αυτά. Ελπίζουμε και η τεχνολογία και η διερμηνία λειτουργήσει καλά. Στις 5.30 θα γίνει αυτό. Όχι σε αυτή την αίθουσα. Στην 4Q1 στο κτίριο Αντάλ Απ' την άλλη μεριά, όπου υπάρχει η τεχνολογία η απαραίτητη, ελπίζω να έρθετε και να συμμετάσχετε, διότι είναι καλή ευκαιρία και σκιώδεις εισηγητές και εισηγητής θα είναι εκεί για να ακούσουν τα όσα θα έχουν να μας πούν οι συνάδελφοι της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως. Και κύριε Σβάμπ, νομίζω ότι έχω δίκιο όταν λέω ότι θα ετοιμάσετε κάποια άλλη δημόσια εκδήλωση ή ακρόαση ανάλογα με την εξέλιξη του κειμένου. Θα υπάρχουν και άλλε ευκαιρίε για συζήτηση. Έχουμε δεύτερη εκρόαση για συμμετοχή εθνικών βουλευτών μετά από αυτή που θα γίνει με τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ε, υπάρχει πολλή δουλειά, πρέπει να γίνει. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την Προεδρία. Το καλωσορίζουμε το εκπρόσωπο εδώ και η κυρία Ρέντινγκ θα προσκληθεί να έρθει το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα προχωρήσουμε το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξη σημαντική γνωμοδότηση για πολιτική ανταγωνισμού. Ελπίζω πολλοί από εσά να μείνετε, διότι ο συγγητής μα, ο κ. Μπίλαν είναι εδώ για να αναφερθεί στο θέμα. Εσείς που δεν θέλετε να μείνετε, αν έχετε την καλοσύνη να αποχωρήσετε σχετικά ήσυχα για να συνεχίσουμε ταχύτερο δυνατόν τις εργασίες μας. Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι το σχέδιο γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής μας για την Επιτροπή Οικονομικών και Μεσματικών Θεμάτων για την ετήσια έκθεση περί πολιτικής ανταγωνισμού. Συντάκτης της γνωμοδοτήσεως είναι ο κ. Άνταμ Μπίλαν και με τα χαράς να του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ο κ. Μπίλαν λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ταχύτητα των εργασιών μας επί της γνωμοδοτήσεως είναι μεγάλη. Αυτό λόγω χρονικών πιέσεων της Επιτροπής Οικονομικών θα προσπαθήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω μάλλον τον πρόεδρο της Επιτροπής και τη Γραμματεία για την απόφαση που ελήφθη για την επόμενη έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο διότι μόνο έτσι μπορούμε να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα για την συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών. Στη γνωμοδότηση εμπεριέχονται 7 σημεία. Στο πρώτο σημείο εκφράζω ικανοποίηση. Καλωσορίζουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο την βελτιστοποίηση της θέσης του καταναλωτού αφιέρωσε ιδιαίτερο ειδικό κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα θέματα των καταναλωτών. Στο δεύτερο σημείο μου αναφέρονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ποια είναι η θέση τους. Το τρίτο σημείο αφορά τη μονάδα διασύνδεσης με τους καταναλωτές της Γενικής Διευθύνσεως ε, Ανταγωνισμού και το διάλογο με τους καταναλωτές ούτως ώστε ε, για να θεσπίζεται η νομοθεσία που αφορά τους καταναλωτές. Το σημείο 4 είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα για τις αποζημιώσεις, για τους μηχανισμούς αποζημιώσεων ε, των θυμάτων παραβιάσεων όσον αφορά τους νόμους αντιτράστ. Αυτό το ζήτημα συχνά το έχει θίξει ο κύριος Σβάμπ. Το θέμα της συλλογικής αποζημιώσεως. Το σημείο 5 αφορά τις ομαδικές εξαιρέσεις που υπόκεινται σε κάθετες συμφωνίες. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα στην Επιτροπή, τα σημεία 6 και 7 σχετίζονται με ομάδες εξαιρέσεων για αυτοκίνητα. Αυτές οι εξαιρέσεις λήγουν φέτος, το Μάιο. Γι' αυτό προτείνω να συμπεριλάβουμε την ημερομηνία 1η Ιουνίου 2010. Δεν μπόρεσα να καλύψω όλες τις προτάσεις των σκιωδών εισηγητών Ελπίζω όμως οι σημαντικότερες προτάσεις ότι έχουν συμπεριληφθεί και αυτό λόγω της ταχύτητας, του ρυθμού που ακολουθούμε, 8 Φεβρουαρίου πρέπει να ψηφίσουμε. Και έχουμε και μεταφράσεις και και γι' αυτό η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι πολύ κοντά. Αύριο στις 12 το μεσημέρι. Λυπούμε γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίλαν που αναφέρατε μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Όπως ξέρετε, για τις γνωμοδοτήσεις δεν έχουμε απεριοριστό χρόνο. Νομίζω όμως ότι κάνατε βέλτιστη χρήση του χρόνου που έχετε και ε, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι θα θέλουν να προσθέσουν κάποια στοιχεία προτού να οριστικοποιήσουμε την έκθεσή σας. Έχουμε τον κύριο Σβάπ, τον ε, κυρία Στάιλερ, τον κύριο Ροσφόρ, ο, κύριε Τριανταφυλλίδη, και εσείς θέλετε να πάρετε το λόγο. Υπάρχει κάποιος άλλος. Η κυρία Τούν είναι εδώ και η κυρία Ράπτη. Δεν ξέρω αν θέλουν ε, να πάρουν το λόγο για να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Δεν θα τους πιέσω όμως. Ε, να δώσω το λόγο στον κύριο Σφάπ, να ε, καλωσορίσω όμως την κυρία Καλούτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σφάπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Μπίλαν για την εξαιρετική του πρόταση. Είναι πράγματι πολύ καλή βάση για την έκθεση στην ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Είμαστε εμείς ε, σκιώδεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα συμβάλλει θετικά στην εκπόνηση της έκθεσης ε, για την πολιτική του ανταγωνισμού 2008. περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη σχέση ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών. Εγώ προσωπικά μία μικρή τροπολογία έχω για το σημείο 4. Επί της αρχής είμαι υπέρ του σημείου 4, απλά θα ήθελα να λέμε ότι τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικούς και και σημαντικούς μηχανισμούς ε, αποζημίωση. και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και τις εργασίες ε, τη επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you Ευχαριστούμε. Κύριε Στάινα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Τα είπε και ο προλαλής σας. Κι εγώ σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Νομίζω ότι είναι συνεκτική. Νομίζω ότι στο σημείο 4 όσον αφορά το θέμα της λογικής αποζημίωσης πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως να προτιμούσα μια διατύπωση που να είναι πιο ισχυρή υπέρ των καταναλωτών. Αλλά έτσι κι αλλιώς πάει προς τη σωστή κατεύθυνση στο σημείο 4. Και για τα 5 και 6 εσείς υπογραμμίζετε το θέμα του κανονισμού για τις εξαιρέσεις είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να δούμε. Με τα καρτέλ, ε, σαν παράδειγμα. όντω πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για το έργο σας και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο με τόσο σφιχτές προθεσμίες. Μέσα σε 24 ώρες πάντως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ροσφόρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μπίλαν και την Επιτροπή για τη δουλειά τους. Μπορώ να πω ότι ο κύριος Σμιτ που μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω γιατί δεν ε, είναι εδώ σήμερα το απόγευμα και αυτός εκτιμά όλος ιδιαίτερος τη δουλειά της Σοφή Χατβέλτ που είναι η από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, εκτιμήσαμε όλους ιδιαίτερος το ότι προσθέσατε μια διάσταση στην οποία αναφερθήκατε και πριν από λίγο για την προσέγγιση υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για μας έχουν τεράστια σημασία. Θέλω εδώ να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Σμίτη και ο και εγώ θα καταθέσουμε τροπολογία ώστε να προσπαθήσουμε να είμαστε κάπως πιο δυνατοί στην προσέγγιση μας υπέρ των συλλογικών αποζημιώσεων. Πιστεύουμε ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να προωθήσουμε το θέμα του ανταγωνισμού. Θέλω να κάνω και μια τελευταία παρατήρηση προς τον εισηγητή. Όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις και τους κανόνες του ανταγωνισμού, εδώ απλά θέλω να πω πως θα θέλαμε τα θέματα αυτά να τα δούμε υπό το πρίσμα του συμφέροντος του καταναλωτή στην Επιτροπή μας. Δεν μπορεί να δείξουμε διαφορία για αυτό το θέμα, τι είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Ροσφόρ. Ο κύριος Τρενταφυλλίδη. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Το μικρόφωνο σας. Επαναλαμβάνω ότι ε, εμείς σαν πολιτική ομάδα ασκούμε κριτική πώς εφαρμόζεται ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά και τι συνέπειες έχει πάνω στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα κάνω πέντε επισημάνσεις κύριε Πρόεδρε για την πολιτική ανταγωνισμού του 2008 και πρώτο σε ό,τι αφορά την επιβολή προστήμου σε καρτέλ. Με την πολιτική επιβολή του προστήμου που ακολουθείται η Επιτροπή πιστεύει πως θα την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης με την νομοθεσία ανταγωνισμού συνολικά. Αυτό όσο και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δεν πάβει να μην είναι επαρκές μέτρο. Απόδειξη συνεχής παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού από εταιρείε κολοσσούς, γεγονό που αποδεικνύει πως το κέρδος είναι μεγαλύτερο από τη δυνητική ζημιά, δηλαδή τον πρόστιμο. Η εκ των υστέρων επιβολή ποινών σε καρτέλ συμπεριφορέ που έχουν σοβαρέ επιπτώσει στους καταναλωτές δεν καθιστά επαρκή θεραπεία αφού κανένας ζημιωθής δεν αποζημιώνεται προσωπικά και έγκαιρα για τη ζημιά που υπέστη, ούτε για τις πιθανές επιπλοκές στην οικονομική του κατάσταση που του προκάλεσε. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, οι πρόσφατες διαπιστώσεις οικονομικών αναλυτών ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει να ξεφεύγει από την κρίση δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει από το γεγονός πως η κρίση ακόμη υποβόσκει μέσα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους πολίτες. Τα μέτρα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν έτσι που να ενισχυθεί η δυνατότητα των κρατών να δίνουν τονωτικές ενέσεις στην οικονομία τους. Σε ό,τι αφορά την αγορά ενέργειας, η πλήρης φιλελευθερωποίηση της αγοράς ενέργειας συνεχίστηκε ακάθεκτα παρά το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν και πάλι ούτε σε αυτό τον τομέα θεσμικά μέτρα εποπτείας της συμπεριφοράς των ιδιωτικών εταιριών ενέργειας που όταν αποκτούν πρόσβαση στα δίκτυα εφαρμόζουν πρακτικές εξόντωσης των δημόσιων εταιριών. Η προνομιακή μεταχείριση του ιδιωτικού τομέα ενέργειας έναντι του δημόσιου μετατρέπει το ίδιο το αγαθό της ενέργειας από δημόσιο σε ιδιωτικό και ως τέτοιο θα πωλείται πολύ πιο ακριβά. Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπήρχε ένα τομέα που είχε αφαιθεί εντελώ χωρί θετικό θεσμικό εποπτικό έλεγχο, ήταν αυτό των τραπεζών. Τέλο, ε, Πρόεδρε, στι τιμέ των τροφίμων, ο μονοπωλιακό έλεγχο των πρώτων υλών από του πολυεθνικού κολοσσού, αλλά και η ολογοπολιακή κατάσταση που επικρατεί στη χοντρική και λιανική αγορά των πρατηρίων πώληση ειδών βασική ανάγκη του καταναλωτή, όπω είναι οι υπεραγορέ, είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της αναξέλεκτης ελεύθερης αγοράς που η Επιτροπή εφαρμόζει με δικά της νομοθετικά μέτρα. Και συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η εφαρμογή του ανταγωνισμού ασθενεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μονόπλευρη εφαρμογή του προ όφελο του ενό κέρδου τη αγορά, δηλαδή τη επιχειρήση, θα πρέπει να αποτελέσει σημείο προβληματισμού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προ αυτή την κατεύθυνση θα είναι και οι τροπολογίε που η δική μου πολιτική ομάδα θα καταθέσει πάνω στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Thank you um, Άλλος κανείς? Ωραία τότε. Η κυρία Σκολούτζη τότε να σχολιάσει αυτά που άκουσε ή ό,τι άλλες παρατηρήσεις έχει να κάνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το κείμενο του κυρίου Βίλαν και για τα σχόλια που ακούστηκαν. Νομίζω ότι είναι επικοδομητικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας βοηθά να ετοιμάσουμε την ε, επόμενη της έκθεση για τον ανταγωνισμό και να τονίσω ότι παίρνουμε στα σοβαρά υπόψη τις απόψεις, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό του 2009. Για τα συγκεκριμένα σχόλια που αναφέρθηκαν, σημειώνω ότι τα ειδικά προβλήματα που είχαμε στους καταναλωτές φαίνεται ότι καλύφθηκαν. Θα το λάβουμε υπόψη στο μέλλον. Υπάρχει ένα πρόβλημα μικροφωνισμού της, από το μικρόφωνο της ομιλήτριας με τα ακουστικά. Καλύτερα τώρα, όχι. Είναι μια προσπάθεια που θα επαναλάβουμε και θα εστιαζόμαστε σε διαφορετικά σημεία κάθε χρόνο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ετέθη το θέμα, να υποβάλουμε πλήρη έκθεση για τη μονάδα σχέσεων με τον καταναλωτή, με τους καταναλωτές. Σωστός διάλογος και διαβούλευση σε θέματα ανταγωνισμού είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και γι' αυτό έχουμε αυτή τη μονάδα για τις σχέσεις με τον καταναλωτή που δημιουργήθηκε το 2008. Αυτή η μονάδα θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με τους καταναλωτές προφανώς αλλά και θέλει αύξηση του διαλόγου με τις οργανώσεις καταναλωτών να παραέχονται απλούστερες σαφείς πληροφορίες προς τους καταναλωτές και το κοινό εν γέννη και πληροφορίες που να είναι σχετικές ε, και να ενημερώνουν τους πολίτες και τους καταναλωτές και ήδη προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκθέσεως αλλά κυρίως την επόμενη έκθεση θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την περιγραφή των δραστηριοτήτων της μονάδας, κάτι που ζητείται από το σχέδιο κειμένου που συζητούμε. Τώρα, λυπάμαι για τους μικροφωνισμούς, λέει η ομιλήτρια. Πιθανόν να πρέπει να χαμηλώσει τα ακουστικά της, την ένταση. I'm almost scared now. <laughs> Φοβάμαι τώρα, εκπέμπω αρνητικά κύματα. Ας προσπαθήσουμε. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις ιδιωτών, είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχετε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα. Καλωσορίζουμε την πρότασή σας και τις τροπολογίες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατα... σχετικά με τη Λευκή Βίβλο υιοθέτησε ένα ψήφισμα το 2009 και εκεί εμπεριείχονται δύο πτυχές που θέλω να τονίσω. χρειαζόταν συνεπής οριζόντια διάσταση προσέγγιση και είναι κάτι που αναφέρθηκε στην έκθεση. Αναφέρθηκε επίσης ότι μια τέτοια συνεπής προσέγγιση δεν αποκλείει την ύπαρξη διαφόρων μέσων. Αυτή η συνέπεια δεν θα πρέπει να επιβραδύνει. Τα τέλεια, τέλεια, το μικρόφωνο δουλεύει. Τη δουλειά, λέω, που γίνεται όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού. Και αυτό είναι κάτι που εμπεριέχεται στο ίδιο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήθελα να επενθυμίσω αυτά τα δύο στοιχεία των συζητήσεων. Για τα άλλα στοιχεία που ετέθησαν όσον αφορά τις κάθετες συμφωνίες, ναι, θα συνεχιστεί ο διάλογός μας με το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό, όπως και με τον κανονισμό για τις εξαιρέσει για τα αυτοκίνητα. Είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο ένα εργαστήριο με το Κοινοβούλιο. Ο διάλογο είναι αρκετά εντατικό και θα συνεχιστεί. Και στην επόμενη έκθεση θα αναφέρονται όλες οι σχετικές δραστηριότητες. Βασικά αυτά ήταν τα λίγα σημεία τα οποία θα ήθελα να θίξω αντιδρώντας τα όσα άκουσα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούσαμε πολύ καλά παρόλο που υπήρχε κάποιο εσωτερικό ανταγωνισμό λόγω ανάδραση με το μικρόφωνο σα, τώρα διθώθηκαν τα πράγματα, υπήρχατε σαφέστατοι. Ο κύριο Μπίλαντ, θέλετε να συνοψίσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα, για τα θερμά τους λόγια, να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας Κατά την εκπόνηση του εγγράφου αυτού δυσκολεύτηκα να συνδυάσω όλες τις θέσεις, όπως για παράδειγμα στο σημείο 4, διότι κάποιες από τις θέσεις σας ε, αποκλείουν η μία την άλλη. Θα εξετάσω όμως τις τροπολογίες και θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο για την ε, ευνοϊκή της νομοδότηση για το έγγραφο αυτό, αλλά και για την υπόσχεση συνεργασίας από την πλευρά της. Ε, και χαίρομαι που μπορώ να σημειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει το διάλογο της ε, με το Κοινοβούλιο για τους δύο σημαντικούς αυτούς κανονισμούς. Να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία, με βοήθησε ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση του εγγράφου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις από την πλευρά μου. Να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι όσον αφορά το θέμα της εξέτασης του Κοινοβουλίου των ε, σχεδίων προτάσεων της Επιτροπής για την αλλαγή των κανόνων ε, για την ε, πώληση και επισκευή μοτοσυκλετών. Η Επιτροπή θα το συζητήσει αυτό αύριο. Ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων μάλλον δεν είναι διατεθειμένη να εκπονήσει έκθεση για το θέμα αυτό. Ίσως να έχουμε προφορική ερώτηση και να καλέσουμε τον αρμόδιο επίτροπο να απαντήσει. Ξέρω ότι θα είσαι εκεί... Ε, αλλά το λέω και για τους άλλους συναδέρφους, διότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να εξετάσουμε και τις τροπολογίες προσεκτικά και να πούμε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ότι αν δεν είναι διατεθειμένη να ασχοληθεί με το θέμα, να μα επιτρέψει εμά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Θα δούμε λοιπόν αύριο τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερον, να επιβεβαιώσω ότι η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι αύριο στι 12 το μεσημέρι. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε λίγο ευέλικτοι, αν πούμε δηλαδή μέχρι το μεσημέρι. Η γραμματεία θα μας επιτρέψει να το ερμηνεύσουμε αυτό με ισπανικό τρόπο. Και να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Μπίλαν, ότι συμφωνήθηκε με τους συντονιστές να γίνει η ειδική συνάντηση στο Στρασβούργο 8 Φεβρουαρίου, Δευτέρα βράδυ, για να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, ώστε να προλάβουμε την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που θα ψηφίσει στις 22 Φεβρουαρίου και ε, στις 2 ε, Μαρτίου θα τεθεί το θέμα στην Ολομέλεια. Έτσι κλείνουμε τις σημερινές μας εργασίες. Να θυμίσω στους συναδέλφους που δεν θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών ότι ε, θα ξανασυναντηθούμε αύριο το απόγευμα στην αίθουσα 4Q1. Παρακαλώ μην αφήσετε έγγραφα στην αίθουσα ετούτη ε, από αυτά που θα χρειαστείτε για την αυριανή συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε με μια ακρόαση με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών. Η κυρία Βάιλερ θα ηγηθεί τη συζήτηση ε, και στι 5.30 ε, θα έχουμε μία ε, βιντεοδιάσκεψη που θα κρατήσει μία ώρα με τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Συνεδρία των συντονιστών αύριο στην αίθουσα τούτη 9 η ώρα το πρωί. Εποφελούμεθα θα έτσι από την ακύρωση τη διάσκεψης των Προέδρων για να κάνουμε προγραμματικές εργασίες. Θα δω λοιπόν του συντονιστέ αύριο. σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή σα. Λήξε τη συνεδρίαση.